Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τι εργασίε μα. αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα. Πρώτο σημείο. χτε έγινε συνεδρία των συντονιστών. Εξετάσαμε όλα τα σημεία της ημερήσιας διάταξης, κυρίως όσον αφορά και το, την ανάθεση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, ενεκρίθη ένα, μια προσέγγιση επανεπολιβουχισμού βάσει της προτάσεως που έκανα ε, το ΑΕΛ και η ΑΛΤΕ. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις θα διανεμηθούν στους συναδέλφους ούτως ώστε όλοι να είναι εν γνώση του συστήματος που θα χρησιμοποιήσουμε το μέλλον, στο μέλλον για να μοιράζουμε γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις όσον αφορά τη διοργάνωση των επισκέψεων και των αποστολών. Ομόφωνα ψηφίστηκε αναβολή της επισκέψεως στην Πολωνία για τον επόμενο χρόνο για λόγους πρακτικούς και πολιτικούς. Επιβεβαιώθηκε και υπογραμμίστηκε, υποστηρίχθηκε η πρόταση της γραμματείας για αποστολή τον Ιούνιο στη Βουλγαρία και διενεμήθηκε το σχέδιο προγράμματος όσον αφορά τις επισκέψεις εις και Ιταλίαν. Θέλαμε να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα και να προγραμματίσουμε τις επισκέψεις μετά τις θερινές ε, διακοπές. Όσον αφορά την Ιταλία, υπήρξε ειδικό αίτημα να συνδυαστεί η επίσκεψη στην Ιταλία, η γνωστή, με την ε, αποστολή την Ελβετική στην Καμπανία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές. Μετά ενεκρίθη και το αίτημα του ΕΛΚ για δύο αποστολές εις Γερμανία. Η πρώτη εις Βερολίνων για συνάντηση με την Bundestag και κάποιους υπουργούς για να συζητηθούν τα θέματα του Jugendamt και μετά να προγραμματίσουμε επίσκεψη για το Σεπτέμβριο στην κάτω Σαξονία, στα σύνορα με Τσεχική Δημοκρατία για να εξεταστούν οι καταγγελίες που έγιναν και συμπεριλαμβάνονται σε κάποιες αναφορές που παραλάβαμε. Το σημείο 3 το θέμα που αφορούσε μια μελέτη για την οδηγία για τα απόβλητα που ανετέθη στη Γενική Διεύθυνση ΠΟΛ. Η μελέτη ενεκρίθη από τους συντονιστές και θα διαβιβαστεί το αίτημα στο Προεδρείο για να προχωρήσει το θέμα γρήγορα. Και σύμφωνα με την πρόταση που έκανε και το Προεδρείο τις περασμένες εβδομάδες. Και συζητήσαμε και την προφορική ερώτηση που πρότεινε ο κύριος Μπουσετήλ με τα τροπολογία στη ΣΑΛΤΕ. και το κείμενο θα δυναμηθεί σε όλα τα μέλη όσον αφορά το θέμα του Ντάμπτ. Ανανεώνεται το θέμα ε, την υποβολή νέων αναφορών. Στη γραμματεία ζητήθηκε να μας δώσει ε, ένα έγγραφο που θα αναφέρει τις αναφορές που έχουν υποβληθεί και τις δρομολογηθήσεις έρευνες για να έχουμε συνοπτική εικόνα των θεμάτων που έχουν τεθεί και να γίνουν τα δέοντα κατά συνέπεια. Τελευταίο σημείο ήταν οι καταγγελίες που ήταν στι αναφορές που υπευλήθησαν από τους πολίτες της αμοχώστου του και κυρίως από την περιοχή των Βαροσίων και να δοθεί συνέχεια στην έκθεση Γκέριγκερ πάνω σε αυτό το θέμα υπό το φως των προσφάτων επισκέψεων που έγιναν μετά από την επίσκεψη του συναδέλφου Βαλέσα και της κυρίας Νεντελτσέβα που την, την περασμένη εβδομάδα υπέσταν και σύλληψη από τις ε, τουρκικές ενόπλες στην νήσο της Κύπρου. Θέλουμε να επαναπρογραμματίσουμε την εξέταση της ε, αναφοράς για να συζητήσουμε το όλο θέμα και μετά να πραγματοποιηθεί μια ερευνητική αποστολή επίσκεψη εις Κύπρον. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδριάσεως, οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ ζήτησαν να την εγκρίνουν γραπτός μέσω ανταλλαγής email δεν ενεκρίθη τις επόμενες ώρες θα εγκριθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 17, το σημείο 17, συνάδελφος Γιάρη το λόγο. Πάρα πολύ σύντομο σχόλιο, Πρόεδρε. Το ε, πρώτο αφορά την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε με τους συναδέλφους συντονιστές για να οργανωθούμε ίσω καλύτερα, γιατί πάντα έχουμε το πρόβλημα ότι η μερίσια διάταξη φτάνει πολύ αργά. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα <clears throat> δεν είναι η αναφορά ΑΟΝΒΕ, αλλά ποιους αναφερομένους θα προσκαλέσουμε, γιατί είναι πολλή δουλειά οργάνωση να έρθουν εδώ και Και μετά έχω πρόβλημα συνείδησης. Όταν τους καλούμε έρχονται και μετά λέμε ότι δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, αισθάνομαι άσχημα. Ε, θα ήθελα να το ξαναδώ με τους συναδέλφους μου και με τη γραμματεία και με ε, την πρόεδρο να βρούμε μία διαδικασία γιατί έτσι πιο μακροπρόθεσμα και πιο οργανωμένα να σχεδιάζουμε ε, τις προσκλήσεις των αναφερομένων. Κάτι άλλο για να μην ξεχαστεί. Είχαμε αποφασίσει στην Επιτροπή μας, ο συνάδελφος Βίλαντ, να κάνει μια προφορική ερώτηση για την Αυστρία. Αν το γράφει αυτό στα πρακτικά ε, και είναι κατοχυρωμένο δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή δεν το ξανασυζητήσαμε χτες τους συντονιστές. Να μην χαθεί, να μην ξεχαστεί αυτό το θέμα για την ε, προφορική ερώτηση για την Αυστρία. Okay. Αυτά. Το είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή, στην Επιτροπή μας αναφορών, όχι στους συντονιστές. Ε, Περδόναμε, Γιάρ. Συγγνώμη, συνάδελφε Γιάρ. Αλλά και έναν των συντονιστών επικρατεί η ομάδα. Εγκρίναμε την πρόταση του συναδέλφου Βίλαν τη συνεδρία τη Επιτροπή και ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα περνά άμεσα στην Ολομέλεια. Δεν χρειάζεται να περάσει από του συντονιστές. Πάμε λοιπόν στο σημείο 17, αναφορά 1447-2009 που υπευλήθη από το Φίλιπ Woolley εν ονόματι της Australian Wildlife Protection Council έχει συλλέξει περίπου 4.000 υπογραφές και αφορά την απαγόρευση εισαγωγή κρέατος και δερμάτων καγκουρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανακοίνωσα χτες, εκείνος που υπέγραψε την αναφορά δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα αλλά είναι εδώ και ο Κρόιτσμαν, εισηγητής της Επιτροπής ΙΜΚΟ, επί του θέματος, που θα αναφερθεί στη θέση της Επιτροπής. Μετά έχουμε παρόντες κάποιους εκπροσώπους της Αυστραλιανής αυτής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Κρόιτσμαν, λοιπόν, έχετε το λόγο. Κύριε Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών μετά από δικό σας αίτημα ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη αναφορά ε, για απαγόρευση εισαγωγής κρέατος και προϊόντων καγκουρό. Και ε, διερευνήσαμε αν χρειάζονται νομοθετικά μέτρα ε, για τέτοιες περιπτώσεις αγωγής κρέατος και άλλων προϊόντων που δεν είναι προϊόντα διατροφής. Στο κρέας κοιτάξαμε τα θέματα της υγιεινής, της ασφάλειας ε, και ε, θεωρήσαμε ότι η Επιτροπή μας δεν είναι αρμόδια για αυτό το θέμα. Η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της ε, αγοράς και δεν χρειάζεται εμείς να δράσουμε. Δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε για το εμπόριο, ούτε ε, φανταζόμαστε ότι θα εμφανιστούν τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Και σύμφωνα με την Επιτροπή μας, σε κανένα κράτος μέλος, κανένα δεν υπάρχουν διατάξεις που να ε, δυσκολεύουν ή να παρεμποδίζουν την εισαγωγή προϊόντων καγκουρό σε όλα τα κράτη-μέλη. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι ε, δεν υπάρχουν πουθενά νομοθετικές ρυθμίσεις. Ξέρουμε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο από πλευράς ε, περιβάλλοντος, αλλά δεν έχει γίνει έρευνα. Οι ε, ε, απαντήσεις των κρατών μελών δεν μας αφήνουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων. Και από πλευράς προστασίας της φύσης επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα. τα είδη καγκουρό που κυνηγούν στην Αυστραλία και παίρνουν τα προϊόντα δεν απειλούνται με εξαφάνιση. Και είναι πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχο και παρακολούθηση από το Μόσπονδα Κρατήδια της Αυστραλίας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε προβλέπονται νομοθετικά μέτρα, ούτε υπάρχουν νομοθετικά μέτρα, ούτε η κοινή γνώμη πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Οπότε από την άποψη της Επιτροπής ΙΜΚΟ δεν χρειάζεται νομοθεσία. Βέβαια, οι επιφυλάξεις αφορούν την προστασία ε, των ζών και είναι κάτι που ξεπερνάει τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Αυτό είναι θέμα που αφορά την Αυστραλία και κατά πόσο η θύρα των καγκουρό ε, είναι κάτι που επηρεάζει ε, την πανίδα εκεί. Ήδη από το 1985 υπάρχει νομοθεσία για την μη απάνθρωπη θανάτωση ε, των καγκουρό, γιατί τα πυροβολούν από απόσταση. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά, προστασία των ζώων στην Αυστραλία, ε, εμπειρογνώμονες που τα κρίνουν και ανθρώπινα και σωστά τα όσα συμβαίνουν. Η Royal Society ε, της ε, Αυστραλίας ε, που είναι μια βασιλική εταιρεία για την πρόληψη ε, των βιωτήτων απέναντι στα ζώα μας απάντησε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο αναφερόμενος τι λέει, ως παραπροϊόν μάλλον η απόρρια και το πρόβλημα, η παράπλευρη η απώλεια είναι ότι όταν κυνηγούν θηλυκά ε, τα ε, μικρά τους, τα ε, μωρά, καγκουρό που είναι έξω από το μάσι που πεθαίνουν γιατί δεν μπορούν να τραφούν. Γι' αυτό μόνο 6 με 8 των περιπτώσεων μάλλον 6-8% των περιπτώσεων αφορά θηλυκά που θανατώνονται. Έτσι λοιπόν, η εισαγωγή αυτών των προϊόντων δεν έχει κανένα πρόβλημα, όχι μόνο από πλευρά εσωτερική αγορά, αλλά και από πλευρά προστασία των ζώων. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν για τη δουλειά που κάνετε και την παρουσία σα εδώ. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λορέντσο Μπονάφο, ο οποίο να εκφράσει την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι υγειονομικέ πτυχέ του θέματο. Κυρία Μπουνάφο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή την απάντηση την έδωσαν οι συνάδελφοι όσον αφορά το θέμα της προστασίας των ζώων και του περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς, θα αναφερθώ στην αναφορά αυτή σε σχέση με το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Ένα μέρος αυτής της αναφοράς αναφέρονται οι συνθήκες υγιεινής, οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές για το κρέας αυτό του καγκουρό γιατί ο χειρισμός του ε, γίνεται μετά από κυνήγι το οποίο γίνεται με οργανωμένο τρόπο. Θέλω να διευκρινίσω, το εξή. όσον αφορά η εισαγωγή ε, κρέατος καγκουρό εγκρίνεται με βάση τον κανονισμό 119 ε, του 2009 όπου καθορίζονται οι συνθήκες εισαγωγής και οι υγειονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρούνται. Όσον αφορά την υπηρεσία επιθεώρησης της Κομισιόν που ονομάζεται Γραφείο Κτηνιατρικών ε, Θεμάτων έγινε ε, μία επιθεώρηση στην Αυστραλία από το γραφείο αυτό με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι συνθήκες παραγωγής αυτού του κρέατος το οποίο εξάγεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται. Στόχος της αποστολής ήταν ευρύτερος βεβαίως από το κρέας καγκουρό αυτό καθεαυτό, όμως μεταξύ άλλων ασχολήθηκαν και με το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας σε σχέση με το κρέας καγκουρό. Τα συμπέρασματα της έκθεσης αυτής είναι ικανοποιητικά. Αναφέρεται ότι οι εγγυήσεις που, που παρέχουν αυτή την εποχή οι Αυστραλιανές αρχές για θέματα υγιεινής είναι ικανοποιητικές. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της προστασίας των ζώων, που εν μέρη κάλυψε ο συνάδελφος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες η Κομισιόν στο θέμα της ευζωίας των ζώων σε ε, τρίτες χώρες και ότι δεν καλύπτεται αυτό το θέμα από τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Επίσης, η Επιτροπή ε, συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αυστραλιανές Αρχές για το θέμα της ε, ευζοίας ε, σε διμερή βάση και ότι υπάρχει κοινή συμφωνία. Ε, το θέμα της ευζοίας προκύπτει συχνά στις επαφές μας με τις Αυστραλιανές αρχές. Εν κατακλείδη, η Κομισιόν θεωρεί ότι η πρόταση που ε, κάνει ο υπογράφων την αναφορά για την απαγόρευση του κρέατος καγκουρό προελεύσεως Αυστραλίας λόγω προβλημάτων πιστιστικής ασφάλειας δεν είναι δικαιολογημένη. Grazie. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια προσέγγιση απόψεων όσον αφορά τα θέματα που εφήγησαν. Χαιρετίζω τον εκπρόσωπο, διπλωματικό εκπρόσωπο της Αυστραλίας, τους εκπροσώπους που είναι εδώ. Επιθυμεί να παρέμβει εκπρόσωπος της Αυστραλίας σε αυτή τη φάση. Αλλιώς να ξεκινήσει τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Τσίτσεστερ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω ως κάποιος ο οποίος ε, είναι επιμακρόν μέλος ε, της ε, κοινοβουλευτικής μας αντιπροσωπείας με την Αυστραλία. Έχω επισκεφθεί τη χώρα επανειλημμένος πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι που με αφορά ε, σε σχέση με το θέμα της αναφοράς. Αγόρασα ένα καπέλο σε μία από αυτές τις επισκέψεις μου που είναι φτιαγμένο από δέρμα καγκούρο. Πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Πρέπει επίσης να πω ότι έχω μεγάλο σεβασμό για, τις, ε, για το ενδιαφέρον των Αυστραλιανών αρχών επί του θέματος. Πιστεύω ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση δεν έχω ιδιαίτερη κατανόηση για αυτή την αναφορά, κυρίως επειδή έχω δεχθεί χωρίς σοβαρό λόγο εξαιρετικά επιθετικό lobbying που φτάνει στο, στα όρια του να είναι και μη ε, Είναι πολύ αντιπαραγωγική όλη αυτή η προσπάθεια. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι από την ΙΜΚΟ και από την Κομισιόν είπαν αυτά που έχουν να πούν. Άρα, εν κατακλείδη, η Επιτροπή μας πρέπει να πει για, το, για την αναφορά αυτή κάτι το οποίο είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τσίτσεστερ. <clears throat> Μια παρατήρηση και μετά μια πρόταση για απόφαση από πλευρά μου. Ε, παρατήρηση πρώτα. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που υπόθηκε. Με το γεγονός δηλαδή ότι η προστασία των ζώων δεν είναι αντικείμενο του ΠΟΕ. Είναι, το γνωρίζω. Και εμείς που ασχολούμαστε με τη γεωργία ε, θυμώνουμε πάρα πολύ, μας εκνευρίζει αυτό το θέμα, γιατί ε, ε, όντως δεν είναι αυτή τη στιγμή εντός του ΠΟΕ, αλλά θέλουμε να τα καλύπτεται, γιατί εισάγουμε τρόφιμα και ε, ζωικής προέλευσης και θέλουμε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Ο κύριος Κρόιτσμαν είχε την καλοσύνη να μην ασχοληθεί μόνο με την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και με την προστασία των ζώων, αν κατάλαβα καλά, και ε, το δικαίωμα στο κυνήγι του καγκουρό. Μπορούμε να απαντήσουμε στην αναφορά και μπορούμε για να την κλείσουμε επίσης και να διαβιβάσουμε στον αναφερόμενο ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το αίτημα του. Αν δεν επιθυμεί να παρέμβει άλλος, οι απόψεις που εξεφράστησαν εκάλυψαν το θέμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έκλεισε αναφορά. Έχουν ικανοποιηθεί όλοι Ικανοποιήθηκαν στι εξηγήσει που δόθηκαν. Ευχαριστώ τον κύριο Κρόιτσμαν για την παρουσία του, για τη δουλειά του και τον εκπρόσωπο της Αυστραλιανής Αρμόδιας Αρχής. Πάμε στο σημείο 18 της ημερησία διατάξεως. Έχουμε την αναφορά 305 του 2010 της Κάρολα Τουαρντέλα. Δεν είναι εδώ η αναφέρουσα. Δίνω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σεμπαστιαν Γκούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με δύο λόγια θα αναφερθώ στο θέμα της αναφοράς αυτής η οποία θέτει τρία θέματα. Πρώτον, τίθεται το θέμα της έγκρισης της ε, καλλιέργειας ε, γεωμήλων αμφλόρα. Η άδεια αυτή χορηγήθηκε στις 2 Μαρτίου του 2010 με σκοπό να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Ε, υπάρχει ένα έγγραφο με μορφή ερωτήσεων απαντήσεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και αναφέρονται τα ωφέλη ε, της καλλιέργειας αυτής από το 2006 και επιβεβαιώθηκε η θετική γνώμη της Σουηδίας το 2004. Υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ε, απόφαση. Η Κομισιόν λοιπόν ε, μελέτησε προσεκτικά την κατάσταση κυρίως επειδή τα γιόμιλα αυτά έχουν ένα γονίδιο που τα καθιστά ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Το 2008 ζητήθηκε ε, μια νέα γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ, η οποία το 2009 επανέλαβε την έγκριση του προϊόντος μετά συνεργασία με άλλους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η ΕΜΑ και η ΣΕΝΤΙΣΕ επί τη βάση αυτής της ε, γνωμοδότησης αποφάσισε η Κομισιόν να εγκρίνει την καλλιέργεια αυτή, η οποία ξεκίνησε από το 2010 και θα συνεχιστεί και φέτος σε περιορισμένη κλίμακα, εξ όσων γνωρίζουμε, στη Σουηδία και κατά πάσα πιθανότητα και στη Γερμανία. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την ποικιλία αραβοσίτου που ανέπτυξε η Μονσάντο, ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός, το ΜΟΝ 90, 810, ε, από το 98 μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 150 διαφορετικές ποικιλίε που περιέχουν αυτή τη γενετική τροποποίηση, περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο ε, Σπόρων. Το 2009 αυτός ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός εγκρίθηκε σε πέντε κράτη-μέλη, κυρίως στην Ισπανία, γιατί 80% των καλλιεργουμένων επιφανειών ε, βρίσκονται στην Ισπανία. Έξι κράτη-μέλη ε, υιοθέτησαν ρήτρε ε, ασφαλείας ε, για τον οργανισμό αυτό, δηλαδή απογορεύουν την καλλιέργεια η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο απαγορεύουν την καλλιέργεια αυτού του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού στα εδάφη του. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ανανέωσης της έγκρισης αυτού του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Η Κομισιόν πήρε θετική γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ τον Αύγουστο του, 8, του 9 συγγνώμη, και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή μελετά τι βήματα πρέπει να γίνουν για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι Πρόκειται κυρίως για τα θέματα της επιτήρησης ε, ε, του γενετικού τροπο, γενετικά τροποποιημένου αυτοοργανισμού, δηλαδή ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν μετά στο περιβάλλον είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Θέλουμε να ενισχύσουμε το σκέλος αυτό κατά την ανανέωση άδεια αυτού του προϊόντος. Το τρίτο σκέλος της αναφοράς αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις, τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις συμβατικές καλλιέργειες, ε, βιολογικές συμβατικές καλλιέργειες. Η συνύπαρξη, όπως ονομάζεται, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να υπάρχει, είναι κλειδί η δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις αυτές ε, στους τρεις αυτού τύπου καλλιέργεια. Το θέμα της ετικετοθεσίας και της σήμανσης είναι σημαντικό, αλλά βεβαίω πρέπει να προχωρήσουμε από αυτού. Τον Ιούλιο φέτος η Κομισιόν ενέκρινε μια νέα σύσταση για αυτή την συνύπαρξη, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιβλέπουν να εξασφαλίσουν καλύτερα αυτή την ελευθερία επιλογής ανάμεσα στις τρεις αυτές, στα τρία αυτά είδη καλλιεργιών. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Άουκεν. κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα δανέζικα. με που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε καθόλου σε αυτή τη σειρά σκανδάλων που απεκαλύφθη. Η, όλη η δίκηση της ΕΦΣΑ έχει ανθρώπους που έχουν πολύ στενές επαφές και συνδέσμους με, την, με διάφορες, διάφορες όπω όπως είναι η Μονσάντο. Δεν, έγινε, δεν έχουν φύγει καν από τη δίκηση, είναι ακόμα εκεί. και αν δεν πιάνονται υπ' φόρο δεν θεωρείται ότι υπάρχει, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όμως υπάρχουν σαφείς κανόνες. Εάν υπάρχει τέτοια πιθανότητα πρέπει να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν έχουν επαφές με τη βιομηχανία ε, δεν μπορούν να ασκούν αυτά τα καθήκοντα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πέρσι ξέσπασαν σοβαρά σκάνδαλα και έχει εμπλακεί πολύ η ΕΦΣΑ ε, έχει πολύ στενές επαφές με τη βιομηχανία. Στην δική μας επιτροπή θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση παρομοίων θεμάτων. Θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία ΕΦΣΑ να λειτουργεί σωστά, να κριθεί σωστά, ούτως ώστε να την εμπιστευόμαστε, να θεωρήσουμε ότι είναι ανεξάρτητος φορέας και να την εμπιστευόμαστε. Δεν είναι αξιόπιστη όμω αυτή τη φάση. Και μετά θα πρέπει να ζητήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντο να προβεί και αυτή σε μια αξιολόγηση τη ε, ΕΦΣΑ. Και μετά από αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη κατεξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εμεί εδώ στη δική μα Επιτροπή είμαστε η Επιτροπή των Πολιτών. Έχουμε το αξιέπαινο καθήκον να εξασφαλίζουμε την πρόσβαση των πολιτών στο Κοινοβούλιο Μέσο εμών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια, οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν επικρατεί τελικά διαφάνεια. Και στελέχη της ΕΦΣΑ απεκαλύφθη ότι είχαν πολύ στενέ επαφές με την βιομηχανία, όπως με τη Μονσάντο. Πρέπει να πούμε τέρμα, τελεία και παύλα. Φτάνει αυτό. Πρέπει η ΕΦΣΑ να αξιολογηθεί ει βάθο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτού του είδους η αδειοδότηση. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις για να έχουν πρόσβαση οι πολίτες στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Ανησυχούν οι πολίτες. Σειρές, πολλά πολλές καταγγελίες έχουμε λάβει. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποκρίνεται ότι τα πάντα είναι μια χαρά, παρά αυτές τις υποθέσεις που αποκαλύπτονται. Και συνεχίζει σαν να μην τρέχει τίποτα. Πιστεύω κυρία Πρόεδρε ότι θα πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ακούει τι επικρίσει. Πέρσι το 2010 είχαμε σωρία υποθέσεων. Σκάνδαλα επί σκανδάλων. Μια αλληλουχία σκανδάλων διαπιστώναμε ότι συνέβαινε πέρσι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα, δεν ανακάλυψε τίποτα. Εξακολουθεί να εξυπηρετεί τη βιομηχανία. Ελπίζω αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις ανησυχίες των πολιτών και τις έρευνες που διενεργήθησαν. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πει κάτι προς υπεράσπισή της. Αλλά δεν αρκεί να πείτε ότι δεν απεκαλύφθησαν επιτόπου αυτά τα σκάνδαλα επ' αυτοφόρου το ΣΥΠΗΝ. Διότι είναι σαφείς οι κανόνες που έπρεπε να εφαρμοστούν. Πρέπει η ΕΦΣΑ να είναι απόλυτα ανεξάρτητη και δεν υπάρχει ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Αυτό μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Η συζήτηση, όπως προβλεπόταν, επεκτάθηκε και σε θέματα που ετέθησαν με τις επόμενες δύο αναφορές που είναι σχετικές. Ίσως θα ήταν καλύτερο να τις εξετάσουμε όλες μαζί, αλλά είχαμε έτοιμα ε, των αναφερομένων να εξεταστούν ξεχωριστά. Γι' αυτό οργανώσαμε και έτσι τις εργασίες μας. Και η κυρία Άουκεν αναφέρθηκε επί της ουσίας και στις καταγγελίες που περιέχονται στις αναφορές του σημείου 19 που αφορούν τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων και συγκεκριμένο κανονισμό που είναι καθοδόν προς έγκριση. Εγώ θα ήθελα να ακολουθήσω την ημερήσια διάταξη δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία και να κλείσουμε. Για το σημείο 18 λοιπόν, που αφορά συγκεκριμένα την απόφαση να δοθεί άδεια στην ΠΑΣΦ να καλλιεργήσει γεώμηλα και αραβόσιτο γενετικά τροποποιημένα, είχαμε την παρέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, κυρία Άουκεν, δεν μιλούσα μόνο για τη διαφάνεια, λέει η κυρία Άουκεν ήταν και το θέμα της ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία των, ε, για την ασφάλεια των τροφίμων της ΕΦΣΑ. Και αυτή αφορά και τη συγκεκριμένη αναφορά. Αφορά την ευθύνη και την ανικανότητα ε, της ΕΦΣΑ, όχι μόνο τη διαφάνεια. Άρα, ήδη τώρα εδώ είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ασχολούμεθα με το θέμα σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ναι, συμφωνώ λέει ο Πρόεδρος είναι θέματα που αλληλεπικαλύπτονται, συνδέονται. Είναι σχετική η, ανα... παρέμβασή αλλά αφορά περισσότερε άλλε δύο ε, αναφορές. Τέλο πάντων, είναι η άποψη τη συναδέλφου Άοκεν. Ο συνάδελφο Γιάρ έχει το λόγο. Ε, ναι. Θα ήθελα να συμφωνήσω εδώ ρητά με την πρόεδρο. Αυτά που λέει η κυρία και αναφορούν περισσότερο την αναφορά υπαριθμών 19, 18 έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο. Εγώ θα άρχιζα διαφορετικά. Ανεξάρτητα από αν μας αρέσουν τα γενετικά τροποποιημένα, αν είμαστε υπέρ ή κατά, τα εγκρίνουμε ή τα απορρίπτουμε, θα ήθελα να σημειώσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά την άποψή μου, έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία για αυτή την ιστορία. Για τη συνύπαρξη των καλλιεργειών, για τους ελέγχου κτλ. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος, και έρχομαι στη συμβαστική πρόταση τώρα, ότι το σύστημα έχει ένα γενέ λάθος μέσα του. Ε, όλοι εκείνοι που συμμετέχουν στις διαδικασίες, ε, οι πολίτες, ε, οι περιβαλλοντολόγοι, οι πολιτικοί είπανε ω ελάχιστο κοινό παρονομαστή ότι θα χρειαστεί μια ανεξάρτητη αρχή που να τα ελέγχει όλα αυτά και να αποφασίζει για τον κίνδυνο. Υποτίθεται ότι αυτή θα ήταν η ΕΦΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Εγώ όταν ακούω κριτικές προσπαθώ να καταλαβαίνω και τα επιχειρήματά του. Η ΕΦΣΑ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε υποψία από την αρχή, περάνω πάσης υποψίας. Να μην την υποπτεύεται κανείς ε, για λόμπι, για ασκήσεις πίεσης, για μαγειρέματα. Και εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης έρευνας και θα πρέπει να επιτρέπεται η έρευνα και να έχουμε και αξιολόγηση του κινδύνου, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να είναι ανεξάρτητη η ΕΦΣΑ και περάνω πάση υποψίας και αμφιβολίας. Και εδώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με την κυρία Άουκεν, να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Γιατί δεν εξυπηρετούμε ούτε αυτούς που είναι υπέρ της γενετικής τεχνολογίας. Εάν η ΕΦΣΑ βγάζει γνωμοδότηση, ε, η οποία στη συνέχεια ε, αμφισβητείται και προσβάλλεται. Θα το ξαναδούμε στην αναφορά υπαριθμών 19. Για την ΕΦΣΑ υπήρξαν εκεί τίποτα διασυνδέσεις, ε, κάποιες παρατυπίες, πώς μπορούμε στο μέλλον να τα αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Ε, και ακριβώς επειδή πρόκειται η γενετική τεχνολογία και γίνονται μάχες σε χαρακόμματα, ό,τι και να λέει η ΕΦΣΑ όμως, ό,τι και να αποφασίζει, πάντα θα υπάρχει κάποιος που δεν θα είναι ικανοποιημένος. Και αυτός που δεν είναι ικανοποιημένος, πάντα θα ισχυρίζεται ότι ναι, καλά την ξέρουμε και την εύσα τι είναι και από ποιον επηρεάζεται. Γι' αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και εγώ θα είχα την αυθόρμητη ε, πρόταση και συμβιβαστική να κλείσουμε τη 18 και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στη 19 όμως αναφορά για την ΕΦΣΑ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. και ε, για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά γενικά. Εμείς τι θέλησαμε την ΕΦΣΑ, οι πάντες, ως ανεξάρτητη αρχή και τη συστήσαμε και την ιδρύσαμε. Τώρα θα πρέπει όμως από κοινού να φροντίσουμε να μην ε, υπάρχει παραμικρή υποψία. Ε, γιατί έχουμε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και μάχες σφοδρότατες. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Η κυρία Άουκεν. Ε, συγγνώμη. Παρακολούθησα τον συνάδελφο για να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για θέμα για να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Αλλά εδώ στην περίπτωση του Γεωμήλου έχουμε ένα γονίδιο που είναι πραγματικά ανθεκτικό στα αντιβιωτικά. Δεν είναι κάτι το ένα μικρό πραγματάκι, κάτι το αθώο, ένα τίποτα, ένα σήμαντο πράγμα. Έχουμε την αξιολόγηση η οποία εξ ολοκλήρου προέρχεται από την ΕΦΣΑ. Στο διάστημα αυτό της αξιολόγησης από την ΕΦΣΑ έχουμε όλες αυτές τις κατηγορίες κατά της ΕΦΣΑ. Όχι ότι έκαναν τη δουλειά τους με τρόπο σφαλμένο, αλλά η ικανότητά τους τίθεται εν κινδύνο. Δεν χρειάζεται δικαστήριο. Δεν χρειάζεται δικαστής να μας το πει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχουν συμφέροντα, αν υπάρχουν σχέσεις, τότε είναι κατάλληλος. Και η ΕΦΣΑ έχει ισχυρές, βαθιές σχέσεις με, την, με τον κλάδο. Και άρα αυτό το θέμα του γεωμήλου είναι θέμα που προκαλεί υποψίες. Αυτό δεν είναι καθόλου αθώα περίπτωση. Οι άλλες, ναι, αλλά όχι το γεώμηλο άμφορ. Ci sono Άλλος που θέλει το λόγο. Και ο Μπουστινάρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, πρέπει να πω ότι οι αξιολογήσεις δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα και πόρισμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σωστή ανησυχία που επικρατεί. Κοιτάξτε τι γίνεται με το περιβάλλον, κοιτάξτε και την καταστροφή που συμβαίνει τώρα στην Ιαπωνία. Τίθενται δραματικά ζητήματα. Π.χ. όσον αφορά τη χρήση πυρηνική ενέργεια εκεί. Για να αναφερθώ τώρα σε κάποιο στοιχείο τη επικαιρότητα. Για να εξαλείψουμε κάθε υπόνοια ότι τα συμφέροντα των παραγωγών των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, τα συμφέροντα της βιομηχανίας δεν εκπροσωπούνται στην ΕΨΑ, θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε η ΕΨΑ να γίνει μια ανεξάρτητη υπηρεσία, πραγματικά ανεξάρτητος φορέας. Υποστηρίζω αυτά που είπε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Γιάρ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σταθούμε λίγο για την ώρα, να σταματήσει για λίγο η πώληση των προϊόντων που δημιουργούν τέτοιες ανησυχίες. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται, πολύ μεγάλα συμφέροντα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν πρόκειται μόνο για ε, παράνομα συμφέροντα, αλλά υπάρχει, ένα, υπάρχει λογική αμφιβολία όσον αφορά τις συνέπειες που έχουν αυτά τα προϊόντα για τη ζωή των πολιτών. Εμείς θα πρέπει να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει έλεγχος των συνεπειών. Γι' αυτό λοιπόν, από τη μία πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγγυηθούμε ότι είναι ανεξάρτητη η έψα, από την άλλη θα πρέπει να παγώσουμε το εμπόριο, τη διάθεση στο εμπόριο αυτών των προϊόντων. Ας υπάρχουν πιέσεις των λόμπι της βιομηχανίας που είναι πολύ επιθετικά αυτά τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιέσεις για να τα δεχτούμε τα προϊόντα. Γιατί εδώ αν ανοίξουμε αυτό, αν το επιτρέψουμε αυτό είναι σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το, το κουτί της Πανδώρας και να έχουμε ανεξέλεκτες συνέπειες μετά. Διότι Ίσως λόγω ελλείψεως πληροφοριών μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διαπιστώσουμε να συμβαίνει μια νέα τραγωδία. Πάντα αποφύγουμε αυτό. Πρόεδρος, είναι ευαίσθητο το θέμα και γι' αυτό θα ήθελα να μου προτείνουν συνάδελφοι κάποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο κύριος Γιάρ έλεγε ότι θα πρέπει να κλείσουμε ε, αυτή την αναφορά, αυτή την άποψη εξέφραση. Αντίθετα, οι συνάδελφοι Άουκεν και Μποστινάρου έχουν θέση αντίθετη. Έχουμε, εγώ κάνω μια πρόταση. Έχουμε να συζητήσουμε, όπως έλεγα και πριν, άλλες δύο αναφορές. Και για να τελειώσω την πρόταση. Λοιπόν, έλεγα, έχουμε να συζητήσουμε άλλες δύο αναφορές. Που θα αφορούν αυτά τα θέματα και αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Γιάρ και η συνάδελφος κυρία Άουκεν για αυτή την αναφορά. Οπότε ίσως μπορούμε να πάρουμε μια ενιαία απόφαση στο τέλος που αναφορά αφορά και τις τρεις ε, αναφορές. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα σε εκείνο που υπέγραψε τις δύο επόμενες αναφορές που όπως ζητήθηκε όμως θα εξεταστούν ξεχωριστά. Έχουμε τον κύριο Brian Jones για την αναφορά υπαριθμών 813 του κυρίου John Bryan. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω και πάλι το λόγο εδώ. Αυτό αφορά την αναφορά 81308. Ανησυχώ λόγω του ότι το σκέλος των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών της ΕΦΣΑ κάνει συνεχώς ε, ελέγχους χωρίς να υπάρχουν ε, ε, ρήτρε ασφαλείας. Πέρυσι έθεσα τις ανησυχίες μου, αλλά στην απάντησή της η Κομισιόν επανέλαβε τις συνήθεις δηλώσεις της σχετικά με τα πρωτόκολλα και τις αποφάσεις της ΕΦΣΑ. Όταν είπα ότι μπορούσε η κατάσταση να ε, ε, βελτιωθεί και πώς θα γίνει αυτό δεν απήντησε η Επιτροπή. Ως ενδιαφερόμενος πολίτης θεωρώ ότι η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με ε, επικοδομητικό τρόπο στην κριτική και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει τώρα με βάση στοιχεία που θα ε, υποβάλλω. Επισημαίνω ότι το Ευρωβαρόμετρο ε, πρόσφατα έδειξε ότι η ανησυχία για τα γενετικά τροπομένα τρόφιμα έφτασε στο 61%. Επίσης, πέρυσι η αναφορά έφτασε με 2,5 εκατομμύρια περίπου ε, με 1,2 περίπου υπογραφές και, ε, ε, που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο Ντάλι, στον Επίτροπο Ντάλι, ο οποίος δεν έδειξε να ε, ενδιαφέρεται για τα αιτήματα των, διολογημένα αιτήματα των πολιτών. Επίσης, επισημένω, πολλές επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί με δείχνουν στοιχεία. Η ΕΦΣΑ δεν παίρνει υπόψη τις εργασίες αυτές και δεν τις θεωρεί λόγους ανησυχίας και η Κομισιόν μοιάζει ότι αυτή την κατάσταση την αποδέχεται. Υπάρχουν υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα. Πρώτον, η ΕΦΣΑ εξακολουθεί να γνωμοδοτεί θετικά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με βάση μη δοκιμασμένες υποθέσεις και εμπιστευτικά και μη δημοσιευμένα στοιχεία που προσφέρουν οι ετούντες. Οι μελέτες αυτές δεν μπορούν να επαναληφθούν ή να δοκιμαστούν από ανεξάρτητους επιστήμονες και αυτό ε, παραβιάζει τις ε, αρχές της επιστήμης. Η σύνθεση των, ε, του, του σώματος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών της ΕΦΤΑ και η ΕΦΣΑ και τη τη εξακολουθεί να έχει σαφή ε, ε, προτίμηση ε, γέννη προς τον κλάδο και γενικότερα προς την, τον κλάδο των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Η σύγκρουση συμφερόντων συνεπάγε, που περιλαμβάνει και τους, το International Life Sciences Institute και το προσωπικό της ΕΦΣΑ έχει τεκμηριωθεί. Τρίτον, η ΕΦΣΑ εξακολουθεί να μην επιμένει για τα δοκιμές ασφαλείας για το ολόκληρο τροποποιημένο, γενετικά τροποποιημένο φυτό, όπως θα ε, φυτευτεί ή θα καταναλωθεί. Υποθέτει ότι οι υποκατάστατες πρωτεΐνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί ασφάλεια ενός γενετικά τροποποιημένου φυτού και ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ε, σημαντικές συνέργειες ή αν ε, ή απρόβλεπτες παρενέργειες που μπορεί να συμβούν. Ούτε η, ε, τέταρτον, ούτε η ΕΦΣΑ ούτε η Κομισιόν έχουν κάνει το παραμικρό για να βελτιωθεί η ε, δημόσια πρόσβαση στα θέματα, στους φακέλου των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Πέμπτον, η Κομισιόν θεωρεί ότι από τη στιγμή που η ΕΦΣΑ έχει αποφασίσει για την ασφάλεια μιας ποικιλία γενετικά τροποποιημένης, το θέμα τελείωσε. Παρά τα αυτά, η επιστήμη είναι γεμάτη αβεβαιότητε και εξαρτάται από την ανοιχτή έρευνα και τι υποθέσει, οι οποίε δοκιμάζονται και τροποποιούνται. Στην υπόθεση των μελετών για τα γενετικά τροποποιημένοι ε, επιστήμονες που ανακαλύπτουν δύσκολα ε, ε, δύσκολα στοιχεία συνήθως ε, μπαίνουν στο περιθώριο και ε, ε, θεωρούνται κακοί. Άσχετα από τι έχει προκύψει, η ΕΦΣΑ ποτέ δεν άλλαξε τη γνωμοδότησή της. Έκτον, η ΕΦΣΑ εξακολουθεί να, να μην επιμένει ότι όλες οι έρευνες που περιλαμβάνονται στους φακέλους να διεξάγονται τουλάχιστον με τα πρότυπα του κόντεξ. Οι δοκιμές για τις ζωοτροφές με υλικά γενετικά τροποποιημένα είναι πάρα πολύ σύντομες για να έχουμε στοιχεία για τι χρόνιε τοξικέ επιπτώσει. Και ω εκ τούτου ζητώ, επειδή ούτε η ΕΦΣΑ ούτε η Κομισιόν έχουν κάνει κάτι για να αντιμετωπίσουν τι ανησυχίε μου, υποβάλλω στην Κομισιόν στην Επιτροπή μια, για ακόμα μια φορά με κάθε σεβασμό τις εξή προτάσει. Παρακαλώ να, θες, να καταγραφεί ότι το Κοινοβούλιο θα επιμείνει ότι η ΕΦΣΑ θα πρέπει να, να, να μεταρρυθμιστεί για να σταματήσει η, η διακίνηση αυτή και να ε, συμπεριληφθεί μια πολύ ευρύτερη βάση εκπροσώπηση. Δεύτερον, παρακαλούμε να καταγραφεί ότι όλες οι έρευνες που περιλαμβάνονται στα, ε, στις, ε, στους αιτήσεων οφείλουν να είναι διαφανείς, να μπορούν να επαναληφθούν και να επαληθευθούν και ότι οι αιτούντες από το, εδώ και στο εξή θα πρέπει να επιβεβαιώσουν γραπτός όλα αυτά εκ των προτέρων, ότι δηλαδή τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα τους θα γίνουν θα μπορούν να γίνουν ε, συγκρίσιμα. Τρίτον, παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τη μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών στις αξιολογήσεις κινδύνου και να υπενθυμίσετε στην Κομισιόν ότι, δεν, ότι υπάρχει διαφωνία και αβεβαιότητα όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας και την αρχή της ε, πρόληψης, η οποία πρέπει πάντοτε να ε, να, υπάρχει, να την έχουμε κατά νου. Είμαι πολύ ευγνώμων στην Επιτροπή και ζητώ παρακαλώ να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Σας ευχαριστώ. Όμως, αν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα, θα σας παρακαλούσα να μιλήσετε και για τη δεύτερη αναφορά, διότι οι απαντήσεις θα αφορούν και τις δύο αναφορές. Yes, uh, no problem. Uh, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τίτλος αυτής της αναφοράς ε, και ε, το αριθμός της είναι 43610. Εξ ονόματος των 13 επιστημόνων που στην αρχή ε, έθεσαν αυτή την επίσημη καταγγελία πέρσι και πολλών άλλων που την υποστήριξαν ρητά, ευχαριστώ την Επιτροπή για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την υπόθεσή μας. Η προηγούμενη μοναφορά αφορά τη σημερινή αξιολόγηση των ε, ε, γενετικά τροποποιημένων, ενώ ε, η δεύτερη για τη μελλοντική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο του εφαρμοστικού κανονισμού και ο τρόπος με τον οποίο εισήχθη μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Στην αρχή φάνηκε ότι το κείμενο αυτό σχεδιάστηκε για να επιταχυθούν οι διαδικασίες έγκρισης και ρυθμιστικές, ε, απαντώντας στην κατάφορη πίεση της ε, κυβέρνησης των ΗΠΑ και του ΠΟΕ για να υπάρξει ένας εναρμονισμός ή συγχρονισμός, λέει, υποτίθεται εντό εισαγωγικών, ε, κατέρωθεν του Ατλαντικού. Ε, μια σειρά από μέτρα που θα άνοιγαν τον δρόμο για πιο εύκολες και πιο φτηνές ε, αιτήσει προ όφελο των πολυεθνικών εταιριών. Αυτό όμω διακυβεύει και το ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και την υγεία και την ασφάλεια των λαών τη Ευρώπη. Επίση, είχε και ρόλο κλειδί η ΕΦΣΑ και εμεί αντιδρούμε σε αυτό. Υπάρχει μια παλιά παράδοση που λέει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν νομοθετεί κιόλας ε, διατάξεις που καλείται να ε, εφαρμόσει στη συνέχεια. Εδώ γίνεται μια διάκριση μεταξύ soft law και hard law της κρίσης νομοθεσίας και κάποιων ρυθμίσεων ε, που εφαρμόζονται εμείς ε, ανησυχούμε πολύ για το παράρτημα 1 και αυτά σας τα έχουμε αναλύσει στην επιστολή του Φεβρουαρίου του 2010 και ε, τον Απρίλιο του 2010. Παρά τις ε, απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με λεπτομερή υπεράσπιση των θέσεων της ΕΦΣΑ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ξανά και ξανά η ΕΦΣΑ υπεραμεινόμενη τονίζει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διακριτικότητα. Ναι, τι θα πει αυτό, μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους, να προβληθεί με πολλούς τρόπους, ε, ανάλογα ε, με την υποτιθέμενη αντιστοιχεία ε, γενετικά και μη γενετικά τροποποιημένων φυτών. Αυτά όμως που αποφασίζει γίνονται νόμος και εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται από ένα όργανο όπως είναι η ΕΦΣΑ με γνωστή μονομέρεια και υπέρ της βιομηχανίας. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να τα αρνούνται αυτά. Έχω να πω τέσσερα βασικά θέματα. Πρώτον, η ΕΦΣΑ έχει υιοθετήσει την έννοια της συγκριτικής αξιολόγηση ε, ως ε, ουσιαστική αντιστοιχία, ε, συνάφεια και ότι γενικά θεωρείται ασφαλέ. ένα φυτό. Αυτά είναι νοησίες από πλευρά επιστημονική. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ελέγχεται ο κίνδυνος των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και φυτών. Ε, τι θα πει επίσης τυχαία adventitious επιμόλυνση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει την ΕΦΣΑ και θέλει να χαλαρώσει τις ρυθμίσεις και θεωρούμε ότι γενικά έχει εγκαταλείψει την αρχή της προφύλαξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όπως αυτό αναφέρεται ε, στις αντίστοιχες οδηγίες. Την οδηγία 2001 κάθετος 18. Καλούμε την Επιτροπή σας να κοιτάξετε πολύ προσωπικά και αυτά που λέει το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ για οριζόντια διάδοση των γονιδίων μεταξύ των φυτών και ε, Όπω λέει και ο καθηγητής Καράσκο, είναι δραματικέ οι συνέπειε για την υγεία, για το περιβάλλον, αλλά και κοινωνικο οικονομικέ, μετά από εισαγωγή ε, μεταλλαγμένη σόγια στη Νότια Αμερική και αλλού. Σε μη ε, μέλη, αυτή η σόγια καλλιεργείται και στη συνέχεια εισάγεται στην Ένωση. Η ΕΦΣΑ δεν... Ε, σε να ελέγξει ούτε τις άμεσες ούτε τις έμεσες συνέπειες. Έχουν ε, την στρεβλή προσέγγιση και την καθόλου διαιτολογική. Δεν κοιτάζω, δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα. Επίσης, υπάρχουν προτάσεις πρόσφατα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, περιορίζουν την καλλιέργεια. Δεν είναι πρακτικό αυτό που προτείνει οι απαγορεύσει να βασίζουν σε πολιτικέ, κοινωνικέ ή θρησκευτικέ αιτίε. Από τη στιγμή που η Εύσορα όμως βγάζει μια επιστημονική ε, γνωμοδότηση, θεωρούν ότι τα πάντα έχουν λύσει. Μα δεν, ε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η επιστήμη. Υπάρχουν τα υπέρ, κατά. Η κυρία Κορίν λεπάς και οι συνάδελφοί της ε, μιλούν για επιστημονικές αβεβαιότητες και τα κράτη-μέλη μπορεί να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια ή να έχουν αντικρουόμενες απόψεις των επιστημόνων. Ε, ενισχύουμε πάρα πολύ από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4 η Δεκεμβρίου 2008 που είναι στο παράρτημα 2 της παρουσίασης δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί ούτε από την ΕΦΣΑ ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή με την υποστήριξη της ΕΦΣΑ απλώς προσπαθεί να υπονομεύσει ή να ανατρέψει αυτές τις αποφάσεις που έχουν τεράστια σημασία για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Ε, Ευγνωμονώ πολύ την Επιτροπή σα που μου επέτρεψε εξ ονόματο των συναδέλφων μου από άλλα μέρη τη Ευρώπη να παρουσιάσω εδώ την αναφορά αυτή και παρακαλώ ε, τα θέματα αυτά που έθεσα υπόψη να τα εξετάσετε σοβαρά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ που ήσασταν ακριβής ε, και περιεκτικός. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, στον εκπροσώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω διάφορα ονόματα εδώ, από σα ζητώ να πάρετε το λόγο σύμφωνα με την ε, σειρά που έχετε καθορίσει εσείς οι ίδιοι να παρέμβετε ως εκπρόσωποι της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω τις απόψεις Κομισιόν όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους της ΕΦΣΑ κλπ όσον αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και την επανεκτίμησή τους. Η στρατηγική για την αξιολόγηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έχει ε, ε, καθιερωθεί πολύ σωστά σε διεθνές επίπεδο. Ε, υπάρχει, προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι η στρατηγική αυτή την οποία χρησιμοποιεί η ΕΦΣΑ, η οποία ε, έχει και τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Είναι συγκριτική ανάλυση, δηλαδή στην ουσία αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση ενός γενετικά τροποποιημένου αραβόστου η μελέτη συγκρίνεται, ε, στηρίζεται στη σύγκριση του γενετικά τροποποιημένου με τον μη γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. Ε, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν όλες οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά φυτά και κατόπιν η έρευνα επικεντρώνεται στο σύνολο αυτών των διαφορών, σε κάθε μία από αυτές τις διαφορές, σε επίπεδο τοξικολογικό, διατροφικό, υγείας κτλ, τα οποία ε, μελετώνται λεπτομερώς. Πρόκειται για μια ε, σωστή επιστημονική προσέγγιση. Οι λεπτομέρειες της προσέγγισης αυτής και το σύνολο όλων των δοκιμών πράγματι αποτελούν αντικείμενο συζήτηση αυτή τη στιγμή μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών με την υποστήριξη της ΕΦΣΑ ώστε να ε, διατυπωθεί ένας κανονισμός που θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται από τους, ε, αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για έγκριση. Αυτό βεβαίως ενισχύει τις ε, απαιτήσει ε, που υπάρχουν για ε, τους ετούντες. ζητών ε, πιο συγκεκριμένα πρωτόκολλα αναλύσεων που πρέπει να πραγματοποιούνται, είτε με αναφορά στα υφιστάμενα πρωτόκολλα, αλλά μετά από άλλη αίτηση θα πρέπει η ΕΦΣΑ να συντάξει νέα πρωτόκολλα, γιατί κάποια πρωτόκολλα σε διεθνές επίπεδο δεν υφίστανται και ζητάμε από την ΕΦΣΑ να τα δημιουργήσει. Αυτό αφορά την οργάνωση των δοκιμών στο πεδίο και τις αναλύσεις. Επίσης, μελέτες ε, τοξικότητας επί 90 ε, ε, ημερών σε ποντίκια. Όσον αφορά την ΕΦΣΑ. Ήρθαμε σε επαφή με την ομάδα η οποία ε, συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους και αυτή τη στιγμή συζητούμε με τα κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη που στηρίζονται από τις Εθνικές Επιτροπές τους και τους επιστήμονες των επιτροπών αυτών και που συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις για να ε, γίνουν αυτές οι ε, επιστημονικές συζητήσεις. Un second point sur lequel je euh, ε, θέλω να αναφερθώ επίσης στην πρόσβαση που έχει, έχει το κοινό στις μελέτες για την αξιολόγηση κινδύνου. Καταρχήν, το σύνολο των φακέλων και με το εμπιστευτικό και με το μη εμπιστευτικό κομμάτι τους είναι προσβάσιμη μέσω ΕΦΣΑ, αλλά και στα 27 κράτη-μέλη, των οποίων ε, οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση. Αυτό είναι ζωτική σημασία για την αξιολόγηση, δεδομένου ότι η ΕΦΣΑ διαβουλεύεται ε, ε, από την αρχή κάθε αξιολόγησης με όλα τα κράτη-μέλη για να γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων. Η διαφάνεια της διαδικασίας εξασφαλίζεται μέσω ενός παραρτήματος όπου υπάρχουν τα σχόλια που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη για τον κάθε φορά υποανάλυση, υπομελέτη, γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Στη διαδικασία έγκρισης πρέπει να επισημανθεί ότι μόλις ε, δημοσιευθεί η μελέτη της ΕΦΣΑ, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν σχόλια επιστημονικού επίπεδου. Εμείς ε, ως Κομισιόν ε, ζητάμε από την ΕΦΣΑ να σχολιάσει αυτά τα στοιχεία. Τα, τα σχόλια αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΑ και άρα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται. Πράγματι ισχύει ότι είναι μεγάλο το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και θέλω να επισημάνω ότι αύριο η Κομισιόν οργανώνει μια συζήτηση και για την ανεξαρτησία αλλά και για τη διαφάνεια της αξιολόγησης κινδύνου αλλά επίσης και για αυτό το σχέδιο κανονισμού της αξιολόγησης των τροφίμων όπως επίσης και για την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Αύριο θα γίνει αυτή η συζήτηση που οργανώνει η Κομισιόν, η οποία θα αναμεταδοθεί μέσω του διαδικτύου. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία που αφορούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτούς καθεαυτούς. Τώρα δίνω το λόγο στους αδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΦΣΑ και τα διάφορα, τις διάφορες επιστημονικές επιτροπές τα πάνελ. Να υπενθυμίσω εν συντομία το πώς δημιουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάμε στον κανονισμό 178, τον ιδρυτικό ε, κανονισμό για την ΕΦΣΑ. Βασίζεται σε διαγωνισμό ανοιχτό και επευλήσαν αιτήσει. Γίνεται πρώτη επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των υποψηφίων με παρατηρητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γίνεται ένα πρώτο κατάλογος ονομάτων που στέλνεται στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχετε στη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να διοριστούν τα μέλη του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στον κανονισμό 178 όπως προανέφερα. Κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτός ο κανονισμός επίσης προ όσον αφορά τα συμφέροντα των μελών προβλέπει μέλη που ξέρουν τι γίνεται στους καταναλωτές, τα συμφέροντα της βιομηχανίας τροφίμων. Άρα απαιτείται να ξέρουν για τη βιομηχανία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και για να υπάρχει αντιστάθμιση, για αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σύστημα δηλώσεων συμφερόντων, συγκρούσεων συμφερόντων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΑ τις δηλώσεις συμφέροντος. Πρέπει να κάνει μια διάκριση μεταξύ συμφερόντων και συγκρούσεως συμφερόντων. Χωρίς συμφέροντα, ο κόσμος δεν έχει γνώση. Είναι προαπαιτούμενο για τη γνώση των συμφέρον. Βέβαια το συμφέρον που προχωρήσει πολύ μακριά και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Άρα υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ συμφερόντων και συγκρούσεως συμφερόντων. Κάτι αναφέρθηκε για, τα, για τις επιτροπές, τα πάνελ της ΕΦΣΑ. Η διαδικασία ακολουθείται και για τα πάνελ. Υπάρχει ένα γενικό σύστημα που αφορά τις δηλώσεις συμφερόντων και τη σύγκρουση των συμφερόντων. Η ΕΦΣΑ έχει ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα για αυτό το θέμα. Για τα μέλη των επιτροπών, των πάνελ, Έχουμε 10 πάνελ, ένα από αυτά αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Για τα πάνελ λοιπόν, στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΑ υπάρχει βιβλιογραφία του κάθε μέλους και οι δηλώσεις συμφερόντων τους. Άρα υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Και ακολουθεί τη διαδικασία όπως η προαναφερθήσα. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι σημαντικότατη η πτυχή αυτή παρά το ότι είχε αυστηρό σύστημα η ΕΦΣΑ ελέγχου συγκρούσεων συμφερόντων, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ότι πρέπει να έχετε σε επαφή με τους φορείς αυτούς, με τις υπηρεσίες αυτές, για να ενισχυθεί περαιτέρω η διαδικασία η προναφερθήσα. όσον αφορά αυτό το σύστημα εναλλαγής. Δηλαδή, προσωπικό, να υπάρχει κυκλοφορία προσωπικό, που υπάρχει κυκλοφορία προσωπικό από τη βιομηχανία προς την ΕΦΣΑ και Τούμπαλιν και αντιστρόφως. Το προσωπικό της ΕΦΣΑ συμμορφώνεται με τους ίδιους κανονισμούς όπως και ε, το προσωπικό των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και εργάζονται σε τομείς όπου μπορεί να συγκρούονται με τα πρώτερα καθήκοντά τους. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και για τις υπηρεσίες αυτές όπως και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι κάλυψε αυτά που υπόθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το προσωπικό εν γέννη και για τα πάνελ της Επιτροπές της Επιστημονικές της ΕΦΣΑ. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο λέει η Πρόεδρος, η κυρία Άουκεν λοιπόν. Λέει... Διερωτώ με τι είδους ε, χάπια παίρνετε στην Κομισιόν και τι αποτελεσματικό τι αποτελεσματικότητα έχουν για να μην καταλαβαίνετε ότι η σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει εκεί, σαφής. Δεν χρειάζεται δικαστήριο για να αποκαλυφθεί η κατάσταση αυτή. Το, το αξιοπρεπέστερο το άτομο μπορεί να είναι ακατάλληλο. Και όταν πηγαίνει κανείς σε αυτούς τους χώρους είναι ακατάλληλος. Όταν αναφέρεται ότι ότι υπάρχει αυτή η διαπλοκή, αυτές η συνεχής επαφή. Το 2008 η Susie Ράιτενς, επικεφαλής της ΕΦΣΑ, πήγε ε, σε εταιρεία κατευθείαν. Χωρίς το παραμικρό ε, έτοιμα να μείνει εκτός του θέματος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ανακαλύφθηκε το Σεπτέμβριο η Νταϊάννα, η επικεφαλής του Συμβουλίου της ΕΦΣΑ, Νταϊάννα Πανάτσι, είχε ευρύς δεσμούς με την βιομηχανία τροφίμων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και μπορεί να είναι αξιόλογα άτομα, αλλά δεν το γνωρίζουμε δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και ελπίζω να μην είμαστε σε περίπτωση μπανανίας εδώ. Η Γερμανία είναι απόλυτα σαφή στην νομοθεσία της. Μόνο σε μπανανίες μπορεί κανείς να πει «Α, ναι, ξέρετε, είναι καλοί οι άνθρωποι αυτοί, οι αξιοπρεπείς και κάνουν αυτό». Όχι, δεν, ναι, δεν, δεν είναι εδώ το ζήτημα. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτές οι... Ε, αναφορές πρέπει να ξεκαθαριστούν απόλυτα. Να πρέπει να, να σταματήσει προσωρινά όλο το σύστημα ε, αδειοδότησης, να σταματήσει προσωρινά, δεν λέω να σταματήσει για πάντα. Η Μονσάντο, ας πούμε, πριν από έξι μήνες έδειξε ότι ε, όσον αφορά τον αραβόσιτο, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται δραματικά, θεαματικά, γιατί οι επιπτώσεις του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού δεν είναι σταθερές. Και αυτό που ονομάζεται monster weed. Α, βγαίνανε διάφορα ε, ζυζάνια τέρατα, monster weeds, δεξιά και αριστερά. Και δεν μπορούσε κανείς να τα αντιμετωπίσει. Φυσικά ε, μετα, μεταβιβάζονται αυτά στην Δανία έχουμε ξεκάθαρη νομοθεσία, αλλά πρέπει να παραμείνουν αυτά σε κλειστό χώρο και μετά να έχουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα στο σύστημα. Κάθε φορά που βγάζουμε αυτές τις καλλιέργειες έξω, κάνουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχω εδώ ένα, πολλά σκάνδαλα, θα το ονόμαζα σκάνδαλα σαφώς, εν εξελίξει. Ακόμα κι αν η ε, Κομισιόν πιστεύει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο καλοί και αξιοπρεπείς και είναι καθαρά τα πουκάμισά τους κλπ. κλπ. Έχουν όμως βαθιά εμπλοκή σε αυτά εδώ. Πρέπει το θέμα να το λύσουμε εδώ και μετά πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις ε, ε, εκ παραχωρήσεως ε, της εξουσιοδότης πράξης για να προχωρήσει. To reality, <clears throat> when we ask, especially the council, but sometimes the commission. Ε, όλο αυτό το ενδιαφέρον που έχουμε να καλούμε ανθρώπους να συμμετάσχουν σταματά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια, αξιόπιστη και να δημιουργεί εμπιστοσύνη σε αυτά που γίνονται στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Evans. Evans. Κύριε Evans έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι ο Δόκτωρ Brian John, ε, παρουσίασε πολύ σωστά την ε, όλη κατάσταση, έκανε σαφείς συστάσεις για το τι θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή εκπροσωπεί ένα ανευρύτατο τομέα της κοινή γνώμης. Και ξέρω και θα συμφωνούν οι συνάδελφοι ότι είναι από τα θέματα που ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες. Εκατοντάδες επιστολών λαμβάνω όσον αφορά το θέμα. Και όπως είπε και ο αναφέρον, η πιο πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξε ότι 61% των Ευρωπαίων είναι αντίθετοι προς την ανάπτυξη τροφίμων, την παραγωγή τροφίμων, γενικά τροφίμων οργανισμών, 59% πιστεύουν ότι δεν είναι ασφαλές τρόφιμο για την οικογένειά τους και ε, έγινε, ζητήθηκε να απαγορευτούν οι καλλιέργειες αυτών των προϊόντων μέχρι να είμαστε σίγουροι τα αποτελέσματα και συνελέγησαν ένα εκατομμύριο υπογραφέ σε αυτό το αίτημα. Αυτό συζητούμε, ένα θέμα που απασχολεί όλες ιδιαίτερα τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε. Να πω δύο πράγματα, διότι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα πιο βασικά Λοιπόν, από τα εξή. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της νομιμότητας της ΕΦΣΑ, κα, κατά πόσο λειτουργεί σωστά. Και δεύτερο, το θέμα κατά πόσο η γνώση που εκφράζεται εκεί είναι ανεξάρτητη επιστημονικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να παρουσιάσει ότι είναι άτομα επιφανή. Αυτό δεν σημαίνει όμω είναι αξιόπιστα σχετικά με αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ότι αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ προσεκτικά και δεν νομίζω ότι το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω ότι είναι δεδειγμένο ή υπεύθυνο η ΕΦΣΑ να είναι ο φορέας που παίρνει τελική απόφαση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οι αξιολογήσεις βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις και στοιχεία που υποβάλλουν οι ετούντες. Με άλλα λόγια, η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, οι εταιρείε που παράγουν αυτούς τους οργανισμούς είναι εκείνοι που παρουσιάζουν τις έρευνες και στοιχεία για να αποφασίσει κανείς κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι ανεξάρτητη η έρευνα ειναι ανεξαρτητη ερευνα αυτη που πραγματοποιείται και στην καλύτερη υπόθεση οι εταιρείε που θέλουν να παράγουν τις γενετικά τροπημένους οργανισμούς δεν θα τονίσουν τα προβλήματα που ίσως διαπιστωθούν όταν κάνουν την έρευνα και το ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιείται περαιτέρω το υλικό που έχουν παράγει αυτή στην έρευνά τους δημιουργεί υπόνοιες. Και βέβαια παρουσιάζουν βολικά και θετικά αποτελέσματα εταιρείε που υποβάλλουν στην ΕΦΣΑ. Το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντο στην ΕΦΣΑ. Αναφέρθηκε αρκετά λεπτομερό. Αυτά τα θέματα έχουν τεθεί ήδη στο Κοινοβούλιο οι σχέσει με διάφορε τέτοιε εταιρείε, των μελών τη ΕΦΣΑ με αυτέ τι εταιρείε, και ζητείται να ε, δημιουργηθεί ένα φορέα επιστημονικό ανεξάρτητο πραγματικά για την αξιολόγηση των γενετικά των οργανισμών. Καλά τα είπε η κυρία Όκεν για τι συμπράξει η Επιτροπή μας πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Αυτό που ζητείτε στην αναφορά, τι είναι. Μεταρρύθμιση, βελτίωση της εξολογήσεως κινδύνων, είναι θέματα που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια. Αφορούν ε, ανεξάρτητη και παληθεύσιμη ε, έρευνα. Και από αυτό ο κύριο Μπράιαν Τζον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008 συμφώνησε με όλα αυτά τα σημεία. Δηλαδή ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ο τομέας Και αποφάσει του Συμβουλίου είναι προσαρτημένες στην ίδια την αναφορά, στα έγγραφα που διενεμήθησαν στους συναδέλφους. Άρα, θα ζητούσε η Επιτροπή να υποστηρίξει την αναφορά αυτά, να υποστηρίξει τα πολύ σαφή και λογικότατα αιτήματα που υπευλήθησαν, ε, σαφή αιτήματα για δράση που έχουμε μπροστά μας, διότι βλέποντας την ομοθεσία που διέπει τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, υποτίθεται ότι πρέπει να δράσουμε σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης. Αυτό είναι στο επίκεντρο της αναφοράς, αυτή η αρχή. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα αύριο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα αιτήματα για δράση στη συζήτηση αυτή, διότι αυτές είναι ανησυχίες ευρέως διαδεδομένες στην Ευρώπη. Ανησυχίες που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή είναι η δυνατότητα που έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι επ' αυτού εκ μέρους του, του λαού που εκπροσωπούμε και υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Άουκεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ο κ. Γιάρη έχει το λόγο. Έχω δύο παρατηρήσεις και ελπίζω μια καλή διαδικαστική πρόταση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Όκεν που έκανε μια διάκριση όταν μίλησε μεταξύ του ε, ε, κλειστού κυκλώματο, γενετική τεχνολογία σε κλειστή διαδικασία, δεν έχει πρόβλημα με αυτό, και του υπολείπου. Ξέρω και τη συζήτηση. Έχουμε και τη λεγόμενη κόκκινη γενετική τεχνολογία στην ιατρική και τη λευκή που είναι στο εργαστήριο που παράγονται κάποιες βοηθητικές ουσίες για τρόφιμα και έχουμε και την πράσινη γενετική τεχνολογία. Και όταν κάποιο απαιτεί να έχει μια ελεύθερη ζώνη από παντού, να μην υπάρχει πουθενά γενετική τεχνολογία, πρέπει να κλείσουμε και όλα τα φαρμακεία, ξέρετε. Προσοχή λοιπόν εδώ. Εγώ ισχυρίζομαι και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι και πολιτικά και επιστημονικά θα πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε για να αξιολογούμε και να μετράμε τον κίνδυνο της πράσινης γενετικής τεχνολογίας. Άλλες χώρες του κόσμου το πράττουν διαφορετικά αυτό. Αλλά θέλω εγώ να φροντίσουμε η έρευνα και η αξιολόγηση του κινδύνου να παραμένει στην Ευρώπη. Γιατί αν τα απεμπολίσουμε αυτά, άλλες χώρες θα αναλάβουν την ευθύνη αυτή που δεν ξέρω αν είναι τόσο επιμελή στον έλεγχο και τόσο σχολαστική όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε ε, όλη γνώση, ο καθένας στη ζωή του ζει διάφορε ε, ε, δραματικές εμπειρίες. Εγώ το ζήσα στην Αργεντινή αυτό, ε, αποστολή επίσημη του Κοινοβουλίου. Και είτε μας αρέσουν κάποια πράγματα είτε όχι, αυτά θα γίνονται αλλού. Και όταν τους ρώτησα, δεν φοβάστε με τη στρατηγική σας ε, ότι θα χάσετε την ευρωπαϊκή αγορά και μου είπε να τη χάσουμε σιγά την αγορά. Εμάς μας ενδιαφέρει η ασιατική αγορά. Εγώ θέλω να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως και η έρευνα και η εξολόγηση του κινδύνου ακριβώς γιατί δεν τα παίρνουμε αυτά αβίαστα υπόψη. Έχουμε γνώση Βέβαια κάποια επιστημονικά θέματα μα ε, ξεπερνούν. Πρώτον θα πρότεινα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητήσουμε γνωμοδότηση για τι επιμέρου επιτροπέ ε, στη 18 για το περιβάλλον και τη γεωργία. Δεν ξέρω σε ποια επιτροπή πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Στη Επιτροπή Γεωργίας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν ξέρω. Παρακαλώ την Πρόεδρο να μας βοηθήσει εδώ, να μας διαφωτίσει. Για την ΕΦΣΑ, για το, την πολιτική προσωπικού σε ποια επιτροπή του Κοινοβουλίου ανήκει αυτό, από ποιον να ζητήσουμε γνωμοδότηση για την ΕΦΣΑ. Και αντικειμενική όμως, αλλά και ε, να είναι αρμόδια η Επιτροπή καθήλυν. Λοιπόν, να παραμένει ανοιχτή αναφορά να ζητήσουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας, επαναλαμβάνω της Επιτροπής Περιβάλλοντος και μια επιτροπή που δεν ξέρω ποια είναι αυτή, να μας πει για το προσωπικό της ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Γιάρο και Μποστινάρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα, θέλω να πω ότι το πιο επικίνδυνο θα ήταν εμείς οι πολιτικοί να κάνουμε τους δικαστές και τους επιστήμονες. Δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Ούτε δικαστές είμαστε, ούτε επιστήμονες είμαστε. Ξεκινώντας από αυτά που ήδη υπόθηκαν από τους συναδέλφους, αναφέρθηκαν στην αρχή της πρόληψης, το λογικό κίνδυνο, αξιολόγηση κινδύνων. Από όλα αυτά εγώ διαπιστώνω ότι τώρα είμαστε στην αρχή μιας κρίσης διατροφικής παγκόσμιας. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που το δείχνουν αυτό. Από τη μία εμεί προσπαθούμε εδώ να δεχθούμε ότι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να συμβάλλουν για την ώρα στην αύξηση της παραγωγής των τροφίμων και ενδεχομένως εμείς να γίνουμε αντικείμενο πολύ ισχυρών πιέσεων από πλευρά τη βιομηχανία. Αν γίνει αυτό θα ήταν πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, ζητούν οι συνάδελφοι και εμείς ακαιρεότητα, διαφάνεια και σωστή διοντολογία να εφαρμόζονται από την ΕΦΣΑ. Και αυτό θα πρέπει να παγιωθεί και να επιβεβαιωθεί. Αυτό ζητά το Κοινοβούλιο. Ε, και στις είπα και στην Ευρώπη έγιναν μελέτες για τα fast food. Τα fast food διαπιστώθηκε ότι έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία. Αλλά τα λόμπι της βιομηχανίας φρόντισαν ούτως ώστε και η ΕΦΣΑ εν τη σοφία της να επιτρέπει να κυκλοφορούν τέτοια προϊόντα στην αγορά. Με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. Και ο φορολογούμενος πληρώνει για αυτές τις συνέπειες, τις αρνητικές. Και κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Η ανθρωπότητα πέρασε κρίση. Την κρίση διαφόρων ασθενειών, μολυσματικών, τη μόλυνση, την ασθένεια των χείρων κλπ. Και τελικά είδαμε ότι το χοιρινό κρέας τότε, μάλλον σήμερα, ε, ε, πωλείται, και πέρα των ορίων που είχαμε καθορίσει μέσω της αξιολογήσεως των κινδύνων. Δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτη εγγύηση στα όσα υπάρχει κάποια αρρωστιολογία από πλευρά ΕΦΣΑ. Χρειάζεται μεγαλύτερη βεβαιότητα. Και αν δεν υπάρχει βεβαιότητα, χρειάζεται καλύτερη ανάλυση του κινδύνου. Αυτό είναι το ελάχιστο. Πρέπει να προστατευτεί και η ευρωπαϊκή αγορά και οι πολίτες από τους κινδύνους. Τέλος θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές και οι τρεις αναφορές. Θα πρέπει να εξεταστούν ομού. Θα πρέπει να αποσταλούν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Γεωργίας και θα πρέπει να υποβληθεί και προφορική ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο ούτως ώστε να μάθουμε για μία ακόμη φορά μέχρι ποιου σημείου είναι πρόθυμη να κινηθεί και να φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με υπευθυνότητα και, την αναγκαία, και στον αναγκαίο βάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα το οποίο φαίνεται και από τις πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές που συνόδευσαν την υποβολή αναφοράς στον Επίτροπο Ντάλι. Άρα υπάρχει θέμα προσυζήτηση και αναμφισβήτητα δεν μπορούμε εδώ να βρούμε τη λύση. Μπορώ να πω όμως ότι υπάρχει ομοφωνία, ότι δεν θα πρέπει να αρχιοθετηθούν αυτά τα θέματα, διότι υπάρχουν καταγγελίες, βάσιμες καταγγελίες και επειδή το θέμα είναι ανοιχτό και συζητείται γενικώ. Άρα, σωστό και πρέπον εμείς να συμμετάσχουμε στη συζήτηση και να εγγυηθούμε ότι τελικά θα δοθεί μια απάντηση που απαιτούν οι πολίτες από την Επιτροπή μας έγιναν προτάσεις. Μεταξύ αυτών το αίτημα προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος να γνωμοδοτήσει. Ανανεώνουμε το αίτημα προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι ήδη είχαμε καλέσει την Επιτροπή να κάνει κάτι τέτοιο και έχουμε μία απάντηση που έχουμε στους φακέλους μας Διαδικαστικά εξετάστηκε το θέμα σε αυτή την Επιτροπή, αλλά δεν μπήκε στην ουσία. Αλλά επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας απευθυνόμενο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και στην Επιτροπή Γεωργίας θα απευθύνουμε νέο αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες παρεμβάσεις της Επιτροπής αυτής. Θα ζητήσουμε λοιπόν και μία συζήτηση με την Επιτροπή ε, Γεωργίας όπως ζητήθηκε. Να ζητήσουμε και άλλα στοιχεία από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σιωπή ήταν η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, αναφορά που ευλήθη σε αυτούς. Θέλουμε και πιο συγκεκριμένα από τον Επίτροπο κύριο Ντάλι να μας πει τι συγκεκριμένο θα κάνει όσον αφορά συγκεκριμένες καταγγελίες που περιέχονται σε αυτές τις αναφορές ε, που θέτουν κάποια ζητήματα που έχουμε θέσει και εμείς. Θέλουμε διευκρινήσεις σε σχέση με τις απαντήσεις μας έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θεωρούμε ικανοποιητικές όμως αυτές τις απαντήσεις. Το είπατε κι εσείς. Εγώ θα προσέθετα και κάτι άλλο. Απευθυνόμενοι προς την Επιτροπή μας. Και προς την Εύσα μάλλον. Απευθυνόμενοι προς την Εύσα Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που εκφράστηκαν και τα προβλήματα εκφράστηκαν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Εύσα θέλουμε κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Επαφές που ίσως οδηγήσουν σε κάποια χρήσιμη διαλεύκανση χρήσιμη για όλους. Με συμβουλεύει η γραμματεία και σας προτείνω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα να αναζητήσουμε την άποψη και τη ΣΤΟΑ που είναι ο φορέας που εποπτεύει τη δραστηριότητα των υπηρεσιών των οργανισμών. Να ζητήσουμε και από αυτό το φορέα λοιπόν, να στείλουμε σημείωμα και να ζητήσουμε από αυτό το φορέα να ε, συμμετάσχει στην όλη προσπάθεια που έχουμε αποδοθεί. Πιστεύω αυτό είναι πρόγραμμα εργασιών, παραμένουν οι αναφορές άνοικτες και θα κάνουμε αυτά που είπα. Και ελπίζω τελικά να έχουμε μια παραγωγή έργου, να μην παραμείνουμε μόνο σε άσκηση επιχάρτου. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ ιδιαίτερα εκείνον που υπέγραψε την αναφορά και ελπίζω να μπορέσουμε να συμβάλλουμε συγκεκριμένο τρόπο στην όλη προβληματική που έχει τεθεί. Πάμε λοιπόν στο σημείο 20 και στις συγκεκριμένες αναφορές του σημείου αυτού. Έχουν σαν αντικείμενο την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος στη Λεόν και στην Σωρία και Νομανσία, στην Καστίγια η Λεόν. Είναι παρόντες όσοι έκαναν την αναφορά Στη Μαρία Γέσους Περέξ Αγορέτα δίνω το λόγο καταρχήν. Σενιόρα Πρεσιδέντα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που δέχεστε και πάλι για ερώτηση από εμάς και μου δίνετε και πάλι την ευκαιρία να έρθω. Είχα έρθει πριν από δύο χρόνια στην Επιτροπή σας σε σχέση με τα έργα που απειλούσαν το φυσικό τοπίο και τον πολιτισμό της Νουμάνσια και τη πόλη της Σόρια. Τότε είχαμε στείλει μια επιστολή στην Υπουργό, μάλλον έστειλε ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής σας ε, επιστολή ε, στην Υπουργό Πολιτισμού και ζήτησε να το αναλάβει αυτό το θέμα το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας για να ε, προστατεύσει την Ουμάνσια από τις οικιστικές παρεμβάσεις που γίνονται. Αυτά ε, βλέπετε που είναι η Νουμάνσια, η κίτρινη γραμμή γύρω-γύρω είναι το τείχος του Σκυπίωνα, του Αφρικανού ε, και έχει αρχαία επίσης το πράσινο είναι η πόλη του περιβάλλοντος ε, και ε, δίπλα έχει μεζονέτες στο Alto Real, ε, μονοκατοικίες. Και επίσης βλέπετε το λεγόμενο βιομηχανικό πολύγωνο, Σόρια 2, είναι βιομηχανική ζώνη η περιοχή. το δικαστήριο του Μπούργος και το διοικητικό δικαστήριο της Σόρια από το 2009 και μέχρι το 2010 παρέλυσαν την απαλωτρίωση για ε, το Σόρια 2, τη βιομηχανική ζώνη που βλέπετε, ε, και εκεί έχει αρχαία, ε, είναι από την εποχή των Ρωμαίων, από το Σκυπίωνα τον Αφρικανό. Είναι πραγματικά παράλογα αυτά τα πράγματα. Χτίζουν επάνω στο πολιτισμό, στην πολιτιστική κληρονομιά. Η οικογένεια Μαριτσαλάρ ε, προσέφηκε στο δικαστήριο, δικαιώθηκε και σταμάτησαν οι απαλωτριώσεις και οι εργασίες. Ωστόσο, παραμένουν κάποιες δραστηριότητες ε, στο βόρειο-ανατολικό, εκεί που είναι η λεγόμενη πόλη του περιβάλλοντος. Και ε, ο νέος οικισμός με τις μονοκατοικίες αυτές τις μεζονέτες. Ε, αυτό ξεκίνησε με ένα βασιλικό διάταγμα το Μάρτιο του 2007 και αποφασίστηκε να ε, χτιστούν εκεί ε, στο Γκαράι και σε 8 χιλιόμετρα από τη Σόρια αυτά τα οικίματα. Είναι στον ποταμό Ντουέρο μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη ε, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το κράτος, ε, το Βασίλειο της Ισπανίας, 19 Ιουλίου ήδη το 2001. Και σύμφωνα με την Οδηγία 9243 του Συμβουλίου, ε, είναι προστατευόμενη η περιοχή ε, για το μεσογειακό τοπίο και τη βιογεωγραφία της Μεσογείου. Επίσης ε, είναι και ιδιαίτερο το έδαφος και χρειάζεται προστασία εκεί γιατί είναι η όχθη του ποταμού του έρω. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουν στους σκοπούς τους άλλαξαν τους κανόνες που ε, διέπουν το καθεστώς αυτό και το χαρακτήρισαν εντός σχεδίου και ότι μπορεί να οικοδομηθεί. Άρχισε λοιπόν στο Σότο καράι η ε, κατασκευή. Όπως βλέπετε όμως πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που είναι δίπλα στο ποτάμι. Και ε, ε, το έχει δείξει και το Εθνικό Σύστημα Χαρτογράφησης του του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι επίσης χαρακτηρισμένη περιοχή ότι πλημμυρίζει. Και απαγορεύεται η οικοδόμηση παντού όταν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που χτίζουν ε, έχει ήδη πλημμυρίσει. Στη συνέχεια θα σα δείξω περισσότερε λεπτομέρειε στα κτίρια. Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση ε, της περιφέρειας Καστήλη και Λεόν, πρόκειται για ένα γενικό σχέδιο ε, αστικής κατάστασης. Εδώ, καταλαβαίνετε, είναι εικονική απεικόνηση από την Ουμάνσια πώς θα φαίνεται. Πάνω από 560 εκτάρια και 500 εκατομμύρια ευρώ έχουν προβλέψει και αυτό και παραθέτω έχει ε, συνδυάσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με ε, όσο γίνεται μεγαλύτερο σεβασμό με το πολύτιμο περιβάλλον ε, και τον περίγυρο. Αυτά λένε αυτοί που το χτίζουν. Έχουν κόψει άπειρα δέντρα. Έχουν αποξεράνει ε, υγρότοπους έχουν καταστρέψει ε, φωλιές πελαργών, τους έχουν φτιάξει κάτι τεχνητές φωλιές που δεν έχουν καμία σχέση με τον οικότοπο και έχουν βάλει και ένα πλαστικό πελαργό για διαφήμιση. Ε, αυτά είναι τρομερά πράγματα. Έχουν χαράξει νέους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει και φαίνεται σαν να είναι νέα κανάλια άρδευσης και υποτίθεται ότι σέβονται πλήρως ε, το περιβάλλον, την κυκλοφορία, την τοπογραφία, τη βελτίωση της φύτευσης και ενεργειακή ε, απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι τα σπίτια που θα χτίσουν εκεί, που είναι πάνω από 700, θα ε, πρέπει όποιος θα αγοράσει να αγοράσει και ένα ηλεκτρικό λέει αυτοκίνητο για να κινείται σε αυτό που ονομάζεται η πόλη του περιβάλλοντος και υπάρχει και μια, ένας θόλος ενεργειακός, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αριστερά, εκεί που ε, θα είναι τα κτίρια και οι υπηρεσίες και οι, οι εταιρείε. Ε, ε, θα είναι κρυστάλλινα, τσιμέντο και γυαλί και θα φτάνουν περίπου στο ίδιο επίπεδο, να το βλέπετε εδώ, με την πόλη της Νουμάνσια είναι γυαλί και τσιμέντο. Και θέλουν να φτιάξουν και πέντε ε, ε, στις όχθες του ποταμού, από εκεί που πηγάζει ο Ντουέρο μέχρι τις εκβολές του. Και, ε, συγγνώμη, μέχρι τα σύνορα με την Πορτογαλία προφανώς και δεν ξέρουμε τι ε, ποσότητα τσιμέντου και γελιού θα καταναλωθεί εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της περιφέρειας Καστίγια Ελαιών, παρά τις απαγορεύσεις, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, παρά όλα αυτά που σας έχουμε επισυνάψει και τα γνωρίζετε και σας είχα πει και πριν από δύο χρόνια, συνεχίζει το πρόγραμμα αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει σε πολλά άλλα σημεία που έχουν προταθεί, χωρίς να καταστρέφεται το ποτάμι και ε, το τοπίο, και, ε, μάλιστα με τρόπο μη αντίστρεπτο. Και είναι ε, πολύτιμο από πλευράς περιβάλλοντος, πολιτιστικής και της κληρονομιάς. 200 επίσης σπίτια, μονοκατοικίες θα γίνουν εκεί που ήταν ο ρωμαϊκός οικισμός του Άλτο Ρεάλ, στο Γκαράι. Επίσης, ε, αυτό είναι μια απεικόνηση ενός ε, καταβλισμού ε, ρωμαϊκού. Αλλά αυτό δεν μπορείς να κάνεις αρχαιολογικά ποτέ. όταν υπάρχουν αρχαία που δεν έχει γίνει εξκαφή, δεν μπορείς να πας να χτίσεις έναν εικονικό καταβλισμό στρατόπεδο. Κοιτάξτε πώς ήταν το στρατόπεδο των Ρωμαίων. Και δίπλα γύρω-γύρω μόνο κατοικίες, ζωνέτες και ε, ουσιαστικά πάνω από 100 σπίτια. Ε, χίλια, συγγνώμη. Και απευθύνομαι και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α, να, κοιτάξτε πώς προχωρούν τα έργα ε, ε για τις βίλες αυτές. Βλέπετε αυτό το λευκό ε, μονόλιθο, εκεί ο αρχαιολόγος Σούλτεν το έχει βάλει αυτό για να δείξει πού ήταν ο καταβλισμός του Άλτο Ρεάλ, του Σκυπίωνα, του Αφρικανού, που είναι ένα σύνολο ρωμαϊκών καταβλισμών, στρατοπέδων, που είναι αρχαία και προστατευόμενα. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας που με δεχτήκατε και δείξατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτιστική, την αρχαία κληρονομιά, όχι μόνο της Ισπανίας, της Ευρώπης ολόκληρης ευχαριστώ την ε, κυρία ε, Δωνα Μαρία Χεσούς Ρουίθ που είναι ε, η τοπική υπουργό περιβάλλοντος. Δεν βλέπετε εδώ τώρα τον οικισμό Γκαρά είναι πίσω από τα δέντρα. Ευχαριστώ όλους εκείνους που βοήθησαν για να σταματήσουν οι εργασίες και να παραλύσουν θέλαμε να απευθυνθείτε και πάλι στην Υπουργό ε, Πολιτισμού της Ισπανίας, την Τόνια Άγγελες Κοσάλης Σίνδε και την Υπουργό Περιβάλλοντος που είναι η κυρία Ελένα Εσπινόσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Μάγερ. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος ε, Αμάλιο Άλβαρο Ντεμαριτσαλάρ, που είναι το όνομά σας. χωρίς μικρόφωνο. Eh, Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του αδελφού μου Άλβαρο Τεμαριτσαλάρ που επιστρέφει από την Αργεντινή και δεν μπόρεσε να Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 2.144 χρόνια η Νουμάνσια ήταν παράδειγμα ε, ελευθερίας και αξιοπρέπειας ενός ε, λαού που δεν ήθελε να υποταχθεί άδικα. Μετά από 20 χρόνια η Ρώμη έστειλε το Σκυπίωνα των Αφρικανών Αφρικανό, τον νεότερο, για να πατάξει την αντίσταση ε, στην Ιβηρική Χεσόνησο. Και η Νουμάνσια τελικά υπέκυψε, αλλά η Ρώμη αναγνώρισε την αξία και την αδρία αυτού του χωριού χωριού και αυτού του λαού και αυτό ε, είναι μια κληρονομιά που μα έχει έρθει μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό για να καταλάβετε τι σημαίνει νουμάνσια, τι, ε, τι, ε, τι αξία έχει ιστορική, πολιτιστική, αρχαιολογική, ε, επιστημονική, λογοτεχνική. Αυτό ανήκει σε όλου και δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να τα χαλάσουμε αυτά, να καταστρέψουμε την κληρονομιά. Επίση στην Ουμάνσια η Ρώμη για πρώτη φορά στην πολιορκία ε, δοκίμασε μια νέα τακτική, μια νέα στρατηγική και μια νέα γνώση που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κάνει την ε, αυτοκρατορία της. Επίσης, ε, γιατί έχουμε τον Ιανουάριο πρώτο μήνα, ε, διότι εκεί ξεκίνησε αυτό στην Ουμάνσια όταν ε, υπέκυψε στη Ρώμη. Επίσης το 1882 μετά από πρόταση ε, της ε, Ακαδημίας της Ισπανίας των Καλών Τεχνών θεωρήθηκε κληρονομιά. Την έχουν υμνήσει οι βασικοί ποιητές μας, οι βασικοί μας συγγραφείς και στην παγκόσμια λογοτεχνία είναι πραγματικά ε, από τα πιο ε, αντιπροσωπευτικά τοπία στην Ευρώπη. Όταν τα βλέπουμε, ξαναζούμε ε, όλη την ιστορία που έζησαν εκεί πριν από 20 αιώνες. Σταματήσαμε μετά από 7 χρόνια με δικαστικό αγώνα αυτό το πρόγραμμα που καταστρέφει και την ιστορική πόλη της Νομάνσια και ε, το περιβάλλον. Συνεχίζουν όμως μετά το 2009 τα έργα, γιατί δεν ανταποκρίθηκαν στα όσα ζήτησε το κοινοβούλιο σας και τόσα επιστημονικά φόρα της Ισπανίας, ακαδημαϊκά πανεπιστήμια και της Ευρώπης και του κόσμου. Χίλια σπίτια στην Ουμάνσια, οχτώ ε, πύργους από γυαλί και τσιμέντο με ύψος 40 μέτρα. Ε, δύο ε, βιολογικοί καθαρισμοί. Αυτό που υποτίθεται ότι λέγεται πόλη του περιβάλλοντος και ε, άλλα 300 σπίτια κολλημένα πραγματικά στο στρατόπεδο του Σκυπίωνα. Δεν έχουμε μάθει από το παρελθόν, δεν έχουμε μάθει από τα λάθη όπως έχουμε καταστρέψει τόσες άλλες περιοχές. Όλα αυτά τα ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα επαναλαμβάνουμε τον 21ο αιώνα. Όλες αυτές οι αξιοθρύνητες πραγματικά δράσεις ε, συμβαίνουν σε ένα υγροβιότοπο, σε μία κοιλάδα που ε, σειραίων υποταμή του Έρο και Τέρα. Και υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικέ ε, λύσεις. Δεν χρειάζεται να πάνε να το βάλουν πάνω στην ομάσια. Ε, στη Σόρια υπάρχει ε, όλη η τεχνολογία, υπάρχει όλη η υποδομή και ε, επίσης θα εξοικονομήσουμε και πολλά χρήματα σε μια κοιλαδα που ε σειραιων του ερο και τερα και υπαρχουν πολλες αλλες εναλλακτικε λυσεις δεν χρειαζεται να το βαλουν πανω στην ομασια στη σορια υπαρχει ολη η τεχνολογια υπαρχει κρίση. Μεταξύ άλλων υπάρχει εναλλακτική λύση της νέας βιομηχανικής ζώνης, της Όρια, που το λένε Βαλκόρβα και θα μπορούσε ε, και το δημόσιο να συμμετάσχει σε αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και θα πιάσουν και περισσότερο τόπο τα χρήματα ε, χωρίς ε, διασπάθηση, χωρίς κατασπατάληση των χρημάτων. Χρειάζεται πραγματικά μια ελάχιστη κοινή λογική. Απλούστατα δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που συμβαίνουν. Χρειάζεται να ενισχυθεί η Λουμάνση, όχι να καταστραφεί, να αξιοποιηθεί το τουριστικό δυναμικό, το οποίο είναι ανεξάντλητο και μόνιμο και σέβονται και το περιβάλλον. Και τέλος, ε, είναι ο σεβασμός στην ιστορία και η καλύτερη κληρονομιά στα παιδιά μας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ κρίσιμη και πάλι ζητούμε την προστασία και τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κάνει ό,τι μπορεί ε, για να προστατεύσει αυτή την κληρονομιά, την ιστορική, την πολιτιστική και την περιβαλλοντική. Υπάρχει και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Περιβάλλον και γενικά οι στοιχειώδεις κανόνες προστασίας ε, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Το καταφέραμε αυτό ήδη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας βοήθησε ε, σταμάτησαν οι απολωτριώσεις, γιατί είναι παράνομες οι διαδικασίες αυτές και παράνομη η αλλαγή του γενικού ε, οικιστικού σχεδίου. Παρακαλούμε να ζητήσετε περιβαλλοντική μελέτη και γενικά μελέτη για το τοπίο όπως όρισαν και οι δικαστές που σταμάτησαν την οικοδόμηση. Και σας παραπέμπουμε στη Βασιλική Ακαδημία Ιστορίας και Καλών Τεχνών επαναλαμβάνουμε τα αιτήματά μας να κάνει το Κοινοβούλιο ό,τι μπορεί όπως ήδη από το Μάρτιο του 2009 αποφάσισε, έτσι ώστε να ε, γίνουν αλλού αυτές οι παρεμβάσεις και όχι στην Ομάνσια. Είναι κοινή λογική, είναι ιστορία που το επιβάλλουν και ο κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σα ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο τώρα στου βουλευτέ, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Γκονσάλε Τεπά. Η κυρία. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί αναφερόμενοι. Πρέπει να σας πω ότι εγώ θα μιλήσω μόνο εξ ονόματο τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τι αντίστοιχε ε, αναφορέ, τι τρει από το 2008, για διάφορα ε, σχέδια γύρω από την ουμάνσια, όπως και η προφορική ερώτηση ε, του Ντάβιτ Χάμερστάιν το 6192 του 2009. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ε, η λεγόμενη πόλη του περιβάλλοντος ήταν ένα έργο το οποίο ε, το 2007 εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η διαδικασία 2105 στις 15 Ιουνίου 2006 έκλεισε. Γιατί δεν μπορούσαμε να αξιολογήσουμε αν θα είχε ε, σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο νόμος 6-2007, περιφερειακός νόμος ε, της Καστήλης και Λεών, έχει ε, προσβληθεί ως προς τη συνταγματικότητά του με απόφαση που έχει δημοσιευτεί και στο Ισπανικό φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης, στην επίσημη Ισπανική εφημερίδα. Έχουν ε, γίνει ασφαλιστικά μέτρα, έχει σταματήσει η απαλωτρίωση και έχει παραλύσει και το σχέδιο ολόκληρο, όπως είπαν και οι αναφέροντες είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι οι εθνικοί δικαστές είναι τα κανονικά τακτικά όργανα ε, τα οποία είναι αρμόδια για να εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκτυο. δίκαιο. Συγγνώμη. Και αυτή είναι μια πρακτική που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει. Σε περίπτωση που εκρεμεί κάτι στην εθνική δικαιοσύνη, για κάποια ζητήματα για τα οποία έχει δεχτεί καταγγελίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, πρέπει να περιμένει την τελεσίδικη απόφαση. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι αιτιάσεις, ε, αλλά είναι υποθέσεις που, ε, σε έκρεμο δικία judice και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί ούτε να ασχοληθεί καθόλου μέχρι να φτάσει η τελεσίδικη απόφαση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσουμε πρώτα το λόγο τώρα στους βουλευτές, η κυρία Γκουτιάρης Κορτίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Ποιο είναι το πρόβλημα. Και το έχουμε επιτάπητος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια γενική παρατήρηση. Όλη η Ευρώπη και το Κοινοβούλιο το ίδιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υφίστανται τις συνέπειες αυτό, της έλλειψης ορισμού για το πώς θα εκτελεί, πώς θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία για την περιβαλλοντική επίπτωση. Η Ευρώπη πρέπει να σέβεται τις συνθήκες και να εφαρμόζονται οι οδηγίες. Η οδηγία για τις ε, περιβαλλοντικές μελέτες λέει ακριβώς ότι θα πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον και ε, η κληρονομιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρει πώς θα ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες που έχει. Ούτε ξέρει πώς να εφαρμόσει το άρθρο 3 της Συνθήκης Λισαβόνας που ενισχύει ε, τη διατήρηση και την προστασία της κληρονομιάς. Δεν ξέρει η Ευρώπη πώς πρέπει να το κάνει, αλλά πρέπει να μάθει η Ευρώπη πώς να το κάνει αυτό. Και από εδώ από το Κοινοβούλιο εμείς θα πρέπει να δώσουμε κριτήρια για το πώς θα αξιολογείται αυτό και πώς θα ασκείται αυτή η εξουσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι σημαντικό αυτό όμως ω προ την κληρονομιά μας. Διότι υπάρχει το εξή στην Ευρώπη. Αν υπάρχει ένας άξονας που χαρακτηρίζει την ιστορία μας είναι ο αγώνας των λαών για τις ελευθερίες τους. Και από εκεί οι διάφοροι λαοί απέκτησαν την ταυτότητά τους. Στην Ουμάνσια ήταν ένα ολοκαύτωμα ενό ολόκληρου λαού που υποτάχθηκε στη Ρώμη, η οποία Ρώμη μας κατέλαβε και έφερε τα δικά της έθιμα κτλ. Ε, αλλά στην Ουμάνσια συνέβη κάτι που μαθαίνουμε στα βιβλία της ιστορίας, στο δημοτικό, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο βιβλίο. Ε, ε, είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας ε, αξιοσέβαστη και θα πρέπει όλοι να την ε, επισκέπτονται. Αυτό είναι άξονας της ταυτότητάς μας. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική. Μάζα ανθρώπων λαοί ολόκληροι ξεσηκώνονται και ζητούν τη ελευθερία τους. Και από την Επιτροπή αυτή εδώ των αναφορών, δεν ξέρω από αλλού, θα πρέπει να πούμε ότι στον κατάλογο της κληρονομιάς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιους χώρους που λέει πέθαναν για να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Δεν φτάνει να πηγαίνουμε να επισκεφτόμαστε το Auschwitz. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των λαών για την ελευθερία και των νεκρών για την ελευθερία. Για την ευρωπαϊκή ελευθερία. Αυτό είναι σημαντικό για την Ουμάσια. Στη συνέχεια η πολιτική μου ομάδα είναι στην εξουσία και εκεί και υπερασπίζεται κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω τώρα. Και τι μας δείχνει αυτή η περίπτωση. Συμμαχούν διάφορες πολιτικές ομάδες υπέρ της καταστροφής της νομάσια. Αυτό είναι μια νέα αντίληψη περί δασών στην Ευρώπη. Φυτεύουμε σπίτια, την να φυτεύουμε δέντρα. Και τι, δηλαδή τα συμφέροντα είναι πιο σημαντικά από τα ιδανικά. Και αν θέλει το κοινοβούλιο να είναι χώρος ελευθερίας θα πρέπει να συνεχίζει να υπερασπίζεται τα ιδανικά ως ε, σημαία και λάβαρο. Γιατί υπάρχουν και τόποι που είναι ιεροί και είναι και τόποι συμβολικοί. Και θα πρέπει να ε, χαρακτηρίζονται ως ιστορικοί τόποι και τόποι μνήμης. Και δεν είναι ο οικότοπο που προσβάλλεται ή καταστρέφεται. Καταστρέφεται η συλλογική μας μνήμη, ο συλλογικός πολιτισμός. Η κληρονομιά συλλογικό πολιτισμος η είναι και άειλη. Εκεί από κάτω έχει στρατόπεδα των Ρωμαίων. Μπορεί κανείς να τα πιάσει, είναι, είναι απτά, είναι χειροπιαστά, μπορεί να τα περπατήσει. Θα πάμε να χτίσουμε εκεί πάνω. Και επίση έχουμε και μια συλλογική μνήμη που είναι αγαθό κι αυτό, δεν είναι θέμα ε, συμφέροντος. Γι' αυτό λέω ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είναι σκάνδαλο πόσα θέματα κληρονομιά φτάνουν εδώ υπό τη μορφή αναφορών στην Επιτροπή μα. Ακριβώ γιατί η Ευρώπη δεν ξέρει πώ να το διαχειριστεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσά να όχι μόνο παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά να μα πει η Κομισιόν. Έχει τη συνθήκη, ωραία. Τι θα κάνει για να διατηρεί το θέμα της κληρονομιάς. Και γιατί μας στείλανε κάποιον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει και προφορική ερώτηση. Δική μας, βουλευτού. Πού να πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι, σε ποια θηρίδα να απευθύνονται, να πούνε χαίρετε, ήρθα να απευθυνθώ για να μου σώσετε την πολιτιστική κληρονομιά. Δεν ξέρει κανείς ποιον να ρωτήσει. Και το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, το αντιληφθεί. Είναι μία μόνιμη αποσία απάντησης για αυτά τα θέματα της χρονομιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε. Η κυρία Άουκεν. Yes. Thank very much. And also... Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη Χριστίνα Γκουτιέρας Καλύφθηκαν πολλά που ήθελα να πω. Γιατί συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Μεγάλο είναι το πρόβλημα. Είναι η πολιτιστική κληρονομιά που αναφέρεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών. Μέχρι τώρα όμως δεν ελήφθη υπόψη σοβαρά. Ήταν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προβληματισμού. Πώς να το πω. Αν εκλέγει ένα λαό με κυβέρνηση που να καταστρέψει την κληρονομιά του, είναι δικό του πρόβλημα. Αυτή είναι η επικουρικότητα για να το πω άσχημα. Είμαστε υπέρ κάποια ε, αλληλεγγύη ε, επικουρικότητας, αλλά έχουμε και κοινή κληρονομιά. Πήγαμε στην Καμπανία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδαμε μεγάλες χωματερές στην περιοχή ε, του πάρκου του Βεζουβίου. Κοινή κληρονομιά, κοινή ιστορία η περιοχή του Βεζουβίου. Άρα υποστηρίζω αυτά που υπόθηκαν. Να ζητήσουμε βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς βλέπει το πράγμα, ποιες δυνατότητες υπάρχουν για κοινή προστασία των κοινών αξιών. όπως τα περιέγραψε τα θέματα αυτά η κυρία Γκουτιέρε και από την Επιτροπή Πολιτισμού. Να ζητήσουμε να τοποθετηθεί, διότι η Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να το ξέρει το θέμα. Πρέπει να μας βοηθήσει. Επειδή είναι αδύναμες οι οδηγίες, σοβαρά υπόψη έχουμε το πρόβλημα. Και υποστηρίζω ένθερμα το να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Εγώ είμαι από τη Σόρια. Εκεί έχω γεννηθεί. Και παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς εξελίσσονται τα έργα στην πόλη του περιβάλλοντος ε, στον πόλο του Γκαράι. Σημειώνω αυτό που είπε η κυρία Γκουτιέρε. Είμαι ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα τη κληρονομία και τη ιστορική κληρονομιά που είναι η Νουμάνσια και είναι η κληρονομιά όλη τη ανθρωπότητα. και θα πρέπει να το προσέχουμε, να το φροντίζουμε αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να σα μεταφέρω και την ανησυχία τη πολιτική μου ομάδας αλλά και ε, του Δήμου τη Σόρια ε, για τα έργα αυτά τη λεγόμενη πόλη του περιβάλλοντο. Έρχεται να τορπιλήσει το θαυμάσιο τοπίο των ερηπείων στην Ουμάνσια. Κάνουν έργα εκεί σε ένα φυσικό περιβάλλον προστατευόμενο. Θα μπορούσαν να το χτίσουν οπουδήποτε αλλού, γιατί σώνει και καλά στον Καράι. Θα ήθελα όμως να πω κάτι ακόμα. Το είπε και η κυρία Γκουτιέρες. Ανησυχούμε όλοι από τη Σόρια ε, για την εγκατάσταση αυτού του οικισμού ακριβώς εκεί. Έρχεται να διαταράξει και την ηρεμία και τη γαλήνη που πάντα επικρατούσε εκεί στην περιοχή. Να τα πείτε αυτά όμως και στο Δήμο του Γκαράη και στην Υπουργό Περιβάλλοντος για, τοπική, γιατί ο Δήμος είναι δικός σας ο Δήμαρχος του Λαϊκού Κόμματος. Και αν κατάλαβα καλά, το πολύγωνο Σόρια 2 έχει σταματήσει. Αυτή η βιομηχανική ζώνη έχει σταματήσει λόγω ασφαλιστικών μέτρων και δικαστικών αποφάσεων. Ευχαριστώ κύριε Ριγκόγεν. Άλλος κανείς? Ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, τους ε, συντάκτες αναφοράς για τη δυνατότητα που έχουμε να ξανάρθετε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Στην πρώτη συζήτηση ε, μας θορύβησε πρέπει να σας πω εδώ στην Επιτροπή μας. Κατάλαβαν όλες οι πολιτικές ομάδες ότι μια πολιτιστική κληρονομιά σαν αυτή της Νομάνσια θα μπορούσε να ε, υποστεί ζημίες ανεπανόρθωτες. Έχουμε τώρα μια καλή είδηση ότι ένα τμήμα του έργου, ε, η βιομηχανική ζώνη Σόρια 2, έχει σταματήσει. Δικαιώθηκαν λοιπόν οι αναφέροντες και επίσης δικαιώθηκε και η συζήτηση που είχε γίνει τότε στην Επιτροπή μας και πιστεύω ότι είναι επίτευγμα και σας συγχαίρω και συγχαίρω και τις πολιτικές ομάδες γιατί καταφέραμε να σταματήσουμε αυτό το τμήμα του έργου. Τώρα, έχουμε τα σπίτια ε, που χτίζονται εκεί και θα πρέπει και εκεί να στείλουμε αξίζει τον κόπο ένα σαφές μήνυμα. Σας προτείνω καταρχάς να στείλουμε δύο επιστολές στην τοπική Υπουργό Περιβάλλοντος και στο Δήμο, όπου να εκφράζουμε την ανησυχία μας για το έργο αυτό και το σχέδιο. Γιατί κατά την άποψή μας, ακριβώς λόγω ε, του τόπου που έχει επιλεγεί, ε, απειλεί την πολιτιστική κληρονομιά. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Γκουτιέρες ε, και πρότεινε, είναι πάρα πολύ εύστοχα και συμφωνώ απολύτως. Και εγώ ανησυχώ και συμφωνώ με την πρότασή της. Και Εφαρμόζοντας το άρθρο 202 εδάφιο 2 του κανονισμού θα πρότεινα στην Επιτροπή Αναφορών να ε, υποβάλουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος για την Ολομέλεια με απλουστευμένη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα πραγματικό έλλειμμα ως προς τις οδηγίες. Γιατί δεν φαίνεται ακριβώς ποια είναι η προστασία που πρέπει να δίνουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό και επευκαιρία αυτή τη συζήτηση που κάναμε για την Ουμάνσια, που είναι σύμβολο του ευρωπαϊκού ε, πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα μπορούσαμε όλες οι πολιτικές ομάδες της Επιτροπής μας να συντάξουμε, επαναλαμβάνω αυτό το αίτημα για την Ολομέλεια με απλούστευμένη διαδικασία, έτσι ώστε να ειδοποιήσουμε, να κινήσουμε όλα τα θεσμικά όργανα, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να ε, έχουν τέτοια έργα και να προωθούν τέτοια έργα όπου ε, βάζουν και το περιβάλλον πάνω από την πολιτιστική κληρονομιά. Και εκτός από τις επιστολές που θα πρέπει να στείλουμε, θα πρέπει να μελετήσουμε συντονιστές πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το άρθρο του κανονισμού 202.2 επαναλαμβάνω για να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα της κυρίας Γκουτιέρης. Με δύο λόγια. Νομίζω ότι η πρόταση να σταλεί επιστολή ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Γιά. Συμφωνώ για το πρώτο, για τις επιστολές. Για το δεύτερο, για το ψήφισμα θα ήθελα να το συζητήσουμε ξανά στους συντονιστές. Με ηρεμία και σύνεση να το συζητήσουμε, όπως επίσης και το περιεχόμενο της επιστολής. Καταρχήν συμφωνώ, αλλά για το περιεχόμενο της επιστολής να το συζητήσουμε στους συντονιστές και για το θέμα του ψηφίσματος επίσης στην Ολομέλεια. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπε ο Πρόεδρος, έχει σημασία. Η κυρία Κορτίνες. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Όκεν είπε επίση κάτι ενδιαφέρον. Αλλά θέλω να προσθέσω το εξή. Σε τέσσερα άρθρα τα λέει η συνθήκη αυτά της Λισαβόνας. Το ένα και πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 3. Και είναι ένα θέμα οριζόντιο, εγκάρσιο. Γιατί πάντα εδώ είμαστε ε, υπό ε, το μανδύα ε, της επικορικότητας ή τη, μεταμφίεση ε, της επικουρικότητας. Λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσουμε και την νομική επιτροπή, ε, αλλά και την επιτροπή στο σύνολό της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλή ιδέα είναι, αλλά να μπούμε στην ουσία του θέματος για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συνεργαζόμαστε. Δεν είναι επίθεση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι εύκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα να καταλαβαίνει τι εξουσίες έχει και να τις ασκεί με τον τρόπο που πρέπει. Ευχαριστώ. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, σημειώνουμε όλα αυτά. Τα τελευταία που είπατε. Και ε, καταλήγουμε. Ε, μένει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ τους συντάκτες που ήρθαν και τη δυνατότητα που είχαμε όχι μόνο να μελετήσουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά να το γενικεύσουμε για να λύσουμε στην Ευρώπη γενικότερα τα όσα συμβαίνουν. Επίσης, ε, να στείλουμε στην αυτόνομη περιφέρεια την επιστολή αυτή και στο Δήμο της Νουμάνσια και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπε και η κυρία ε, Γουτιέρες γιατί είναι πολύ σημαντικό και στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών να συζητήσουμε την εφαρμογή του άρθρου 202 του δικού μας κανονισμού. Εντάξει, για να ε, εγκρίνει ένα ψήφισμα η Ολομέλεια και να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζήτησε ο κύριος Γιάρ. Ξαναζητήσατε το λόγο. Δεν ξέρω. Μήπως δεν κατάλαβα κάτι καλά από τη μετάφραση. Να δούμε και το, την ουσία, το, το περιεχόμενο των επιστολών που θα στείλουμε, να το συζητήσουμε στους συντονιστές. Όχι απλώ να συζητήσουμε αν θα στείλουμε επιστολές και τι θα λένε. Δεν το άκουσα από τη διερμηνία. Δεν ξέρω αν το είπατε, Πρόεδρε. Συνολιά. Κύριε Γιά, προφανώς. Όλες οι επιστολές είναι στη διάθεση των πολιτικών ομάδων, αλλά η επιστολή θα αντανακλά αυτά που συζητήσαμε εδώ. Ότι ανησυχούμε και θέλουμε να ενημερώσουμε και του αρμοδίου και της αυτόνομης περιφέρειας και του Δήμου. Νομίζω ότι και η, ε, γραμματεία θα το κοιτάξει και θα το στείλει σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Α, συντάκτες της αναφοράς... Ε, ναι, κύριος Δεμαρή Τσαλάρ, θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, με κάθε ταπεινότητα να προτείνουμε να στείλετε και μια επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού, διότι η κυβέρνηση ε, ε, είναι ο βασικός ε, αρμόδιος. Εντάξει, βεβαίως και στην τοπική κυβέρνηση και στο Δήμο Σόρια και στο, στο Δήμαρχο του Γκαράη, αλλά θα παρακαλούσα και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ναι, ναι, είναι εύστοχο αυτό βεβαίως, γιατί ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτά. Είναι ε, αρμοδιότητά της. Καλώς. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο 21. τον Άλβαρο Φερνάντε Δουράν Ισπανική Ιθαγένεια σχετικά με ένα έργο αυτοκινητοδρόμου στα Πυρηναία, στην Ισπανία. Αποσιάζουν οι αναφέροντε. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει ενημερώσει και διαζώσεις και με ανακοινώσεις για το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε ε, για την αναφορά αυτή. Για το αντικείμενο το οποίο έχει να κάνει με ένα έργο αυτοκινητοδρόμου στη Σαραγώσα ε, ε, που συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Α21. Είναι ένα ευρύτερο έργο μεταξύ Χάκα και Ναβάρα. Είναι ο αυτοκινητόδρομος Α21 και εδώ πρόκειται για μια μικρή παράκαμψη, για μια μικρή ε, οδό. Και στα πλαίσια ε, αυτού του έργου, του συνολικού όμως, ε, ελέγξαμε και ερευνήσαμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελικά ε, μπορούμε να πούμε ότι ήδη από το Δεκέμβριο του 2002 συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές ε, του Βασιλείου της Ισπανίας είχαν κάνει μια δήλωση ε, θετική ε, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το διάδρομο αυτό Α21 που διέρχεται από τα Πυρηναία και την περιφέρεια της Αραγωνίας. Έτσι λοιπόν η μελέτη αυτή περιβαλλοντική συνιστά την τελευταία φάση της διαδικασίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή έγινε αξιολόγηση, εκτίμηση του περιβαλλοντικού ε, αντικτύπου για το σχέδιο αυτό, το έργο του αυτοκινητοδρόμου και ήδη από το προπαρασκευαστικό στάδιο μελετήθηκαν 56 εναλλακτικέ λύσεις και 11 πιθανοί διάδρομοι, χάραξη δηλαδή του αυτοκινητοδρόμου. Στη συνέχεια οι 6 από τους 11 αυτοκίνητοδρόμου. Ε, αυτοκινητοδρόμους χωρίστηκαν σε διάφορα τμήματα και πάλι μελετήθηκαν οι εναλλακτικέ λύσεις και ορίστηκαν μέτρα ελαχιστοποίησης ή διόρθωση του αντικτύπου. Και στους οικοτόπου που θα θυγούν και τη χλωρίδα και την πανίδα που υπάρχει εκεί ή που μπορεί να υπάρχει. Με τις εναλλακτικέ λοιπόν επιλογές που έγιναν τα έργα, τα τεχνικά που επελέγησαν και τα μέτρα διόρθωσης που προτάθηκαν, συνέχισε το έργο και δεν αναμενόταν να επηρεάσει σημαντικά ε, τους τόπους ε, και τους οικοτόπους από που ε, περνάει ο αυτοκινητόδρομος. Ήδη στη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου το 2002 υπήρχε και ένας όρος που έλεγε ότι σε περίπτωση τροποποίησης του έργου, ε, ε αν ε, μειωθούν οι ε, περιφέρειες που πλημμυρίζουν, περιοχές που πλημμυρίζουν, γιατί ε, θα μετατραπεί και μια τεχνητή λίμνη, μια, ένας ταμιευτήρας εκεί, θα μπορεί να αλλάξει και πάλι κάποιος σχεδιασμός για να είναι όσο γίνεται μικρότερη η καταστροφή ή η βλάβη για το περιβάλλον. Αυτό ε, και συνέβη. Επανασχεδιάστηκε ε, η λίμνη, η τεχνητή λίμνη, μειώθηκε ο όγκος από 525 σε 510 και ε, ο οργανισμός αυτός που έχει αναλάβει το έργο του αυτοκινητοδρόμου, έκανε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις από το αρχικό έργο και ήταν θετική η ε, αξιολόγηση. Οπότε, αυτό εντάσσεται ε, στο δεύτερο παράρτημα της οδηγίας και το πρώτο παράρτημα επίσης έχει εγκριθεί. Μιλώ για την οδηγία για προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει με μελέτη ε, να ορίζουν κάποια κριτήρια ή κάποια κατόφλια, κάποιες οριακές τιμές, για να δουν από ποιο έργο, από ποιο στάδιο και μετά χρειάζεται τέτοια μελέτη που εμπίπτει από την, στην οδηγία. Και στη συνέχεια υπάρχει και το παράρτημα 3 που ε, έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ε, τη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου, τον αντίκτυπο. Το 2006 αποφασίστηκαν αυτά. Και ε, γίνονται κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές νέες μελέτες, νέες έρευνες. Η τροποποίηση λοιπόν του έργου έχει αξιολογηθεί, έχει μελετηθεί, έχει διερευνηθεί και υποβληθεί σε πλήρη ε, ανάλυση. Συμπέρασμα. Με βάση όλα αυτά που σας είπα, δεν έχει διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θέλει κανείς συνάδελφος στο λόγο. Ε, αν δεν θέλει συνάδελφος στο λόγο, θέλω εγώ να πω το εξής. Uh, Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι η αξιολόγησή της συμφωνεί ότι έγινε σωστή αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών, ότι δεν υπάρχουν σοβαρές συνέπειες όσον αφορά το περιβάλλον από την ε, εφαρμογή και η υλοποίηση του έργου αυτού, εγώ θα έλεγα αυτή η αναφορά να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνοντα υπόψη τα όσα είπε ο κύριο Μποστινάρου, το μόνο που έχω εγώ να σας πω είναι πριν κλείσει αυτή η αναφορά να ζητήσουμε ενημέρωση από τη Γαλλία διότι είναι περίεργη αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε που έχει να κάνει και με ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός φτάνει μέχρι ε, τα Πυρηναία, μέχρι την κορφή των Πυρηναίων στην Ισπανία, αλλά το γαλλικό τμήμα δεν είναι αυτοκινητόδρομος, διότι προστατεύεται η, ε, γαλλική πλαγιά των Πυρηναίων και δεν επιτρέπεται να γίνει αυτοκινητόδρομος. Τα Πυρηναία όμως είναι Πυρηναία και στη Γαλλία και στην Ισπανία τα ίδια. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο έργο όπου στη μία πλαγιά των Πυρηναίων να επιτρέπεται αυτοκινητόδρομος που θα συνδεθεί με τη Γαλλία, αλλά μόλις περάσουν τα σύνορα είναι προστατευόμενη ζώνη και απαγορεύεται ο αυτοκινητόδρομος. Πριν κλείσουμε λοιπόν την αναφορά να ζητήσουμε ενημέρωση από τη Γαλλία για να μας πει η Γαλλία πώς έλυσε το πρόβλημα εκεί και με ποιο κριτήριο. Σε ε, ότι μπορεί να γίνει δρόμος εκεί, αλλά όχι αυτοκινητόδρομο στη Γαλλία. Ε, τι λέτε, να ζητήσουμε επιπλέον ε, ενημέρωση. Thank you. As far as I know... Ευχαριστώ. Εξ όσων γνωρίζω, η μόνη προϋπόθεση για να παράσει μια, ένας αυτοκινητόδρομος στη Μεθόριο είναι είτε το έργο να έχει συμφωνηθεί διμερώς ή να είναι μέρος του TNT, των διευρωπαϊκών αξώνων, που δεν είναι η περίπτωση. Και ρωτάω ε, απευθείας τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ε, εντάσσεται αυτός ο αυτοκινητόδρομος σε κανένα διευρωπαϊκό δίκτυο? Όχι. Αν λοιπόν δεν ε, είναι ούτε κομμάτι του δικτύου, ούτε ε, εντάσσεται σε κάποια διμερή συμφωνία, γιατί να ζητήσουμε από τις ε, αρχές να μας στείλουν επιπλέον πληροφορίες. Δεν θέλω να βαρύνω περισσότερο το ζήτημα, ούτε να ενοχλήσω κανέναν. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα είναι απολύτως σαφή σε σχέση με πολλές άλλες περιπτώσεις που έχουμε και έχουμε ακόμα δύο Ανοιχτέ αναφορές στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι ε, επαναλαμβάνω να, ε, την πρότασή μου να κλείσει αυτή η αναφορά. Η κυρία Άουκεν. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει το εξή. Γιατί από ό,τι άκουσα από τον Βίλι Μάιερ δεν είναι θέμα ότι έχουμε ένα έργο αυτοκινητοδρόμου. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της προστασίας της περιοχής. Αν πρόκειται για πλήρως προστατευόμενη περιοχή στη Γαλλία, με συγχωρείτε, ρωτάω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, να ρωτήσουμε από τους εκπροσώπους της Κομισιόν που παρίστανται, αν έχουν αυτά ληφθεί υπόψη και στη Γαλλία. Γιατί και εκεί υπήρξε μια διαφορετική προσέγγιση για την προστασία των ωραίων αυτών. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco de esto quería... Μάλιστα. Ούτε εγώ θέλω να προκαλέσω κανένα πρόβλημα. Ε, ο κύριο Γιάρ, μια σκέψη έκανα. Ναι. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μποστινάρου. Ούτε αυτό είναι τμήμα της αναφοράς. Η αναφορά περιορίζεται ε, στην πλευρά των Πυρηναίων ε, που βρίσκεται στην επικράτεια της Ισπανίας. Είναι λογική η απάντηση. Αλλά εμείς δεν πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο της αναφοράς. Υποθέτω ότι από τη γαλλική πλευρά δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλιώς θα έχει έρθει και η γαλλική αναφορά. Νομίζω ότι μπορεί να κλείσει η αναφορά αυτή, χρειάζεται να την κρατήσουμε ανοιχτή. Και αν υπάρξει πρόβλημα από την άλλη πλαγιά των Πυρηναίων τη Γαλλική θα το μάθουμε. Αυτό θα ήταν ο σωστός δρόμος. Να μην παίρνουμε τώρα εμεί πρωτοβουλία και ε, διευρύνουμε πάντα το αντικείμενο των αναφορών. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Άρου να κλείσει. Και η απάντηση να θεωρηθεί επαρκής. Ο πρόεδρος. Εντάξει. Θεωρείται λοιπόν ε, ότι κλείνει η αναφορά, ότι έχει διεκπεριωθεί και ως γενική σκέψη το είπα εγώ ότι είναι ενιαία διέρετα τα πυρηναία ευρωπαϊκά βουνά, αλλά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σε δύο γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς κυκλοφορεί κανείς στα πυρηναία. Λοιπόν, 22 είναι του κυρίου Ντανιέλ Εγκομπούρου, γαλλικής ηθαγένειας. Εξ ονόματο των Πρασίνων τη Χώρα των Βάσκων, η οποία συνοδεύεται από τέσσερι υπογραφές σχετικά με το αεροδρόμιο της Φουέντεραμπία. Παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενο, μιλήστε, αλλά όχι πάνω από πέντε λεπτά παρακαλώ. Έχω την τιμή να εμφανίζομαι ενώπιόν σας εξ ονόματο της περιβαλλοντικής οργάνωση. Ε, του βιδασόα που είναι στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας. Έχουμε μαζέψει υπογραφές κατά ενός έργου ε, επέκτασης του διαδρόμου της, ε, του αεροδρομίου του Φουενταραμπία. Πρέπει να γίνει αντιληφθό, αντιληπτό το διακύβευμα από γεωγραφική ε, άποψη. Εδώ είναι ο χώρος, η περιοχή δεξιά, κάτω βλέπετε την πόλη Φονταραμπή 16.000 κατοίκων. Επάνω υπάρχει η πόλη των 60.000 κατοίκων, ερών, και κάτω και αριστερά η πόλη ε, Αντάιχ και η πόλη και η παραλία της πόλης. Υπάρχει το μοναστήρι, ε, ε, ο κόλπος, το υπάρχει και ένας, ε, ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο αυτού του συγκροτήματος της ε, ευρύτερης περιοχής της Φουενταραμπία. Δεν βλέπουμε καλά, αλλά εντελώς αριστερά βλέπετε το αεροσκάφος και ο διάδρομος του αεροδρομίου βρίσκεται εκεί κοντά στο, στην παλιά πόλη της Φουενταραμπία. Και σε, πρώτη, βέβαια, σε πρώτο πλάνο ο κόλπος. Ε, τώρα, ποιο είναι το αντικείμενο της αναφοράς. Η επέκταση του αεροδρομίου θα αυξήσει τους κινδύνους. Θέλουν να αυξηθεί φυσικά ο αριθμός των πτήσεων, γι' αυτό επεκτείνεται ο διάδρομος. Γιατί γιατί θέλει να επεκταθεί ο διάδρομος, γιατί δεν συνάδει με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ποιος είναι λοιπόν αντίθετος σε αυτή την, την ε, επέκταση. Υπάρχει μαζική αντίδραση από πλευράς Γαλλίας. Έχουμε σε μια πόλη 90.000, σε μια ευρύτερη περιοχή 90.000 κατοίκων έχουμε συγκεντρώσει περίπου 20.000 υπογραφές και το Γενικό Συμβούλιο, ο νομάρχης που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, είναι τελείως αντίθετος, όπως και οι τοπικές αρχές, στην επέκταση αυτού του αεροδρομίου. Γιατί υπάρχει αυτή η μαζική αντίδραση, επειδή θα αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο ο αριθμός των οχλήσεων που ήδη υφίστανται. Εδώ υπάρχει μια άλλη άποψη του αεροδρομίου που το βλέπουμε εδώ στο κέντρο. Υπάρχει παραλία του Αντάγη με 3 χιλιόμετρα ε, λεπτής άμμου ε, στον κόλπο βλέπετε την ίσο των πουλιών που είναι ακριβώς στον άξονα του αεροδρομίου και εδώ βλέπετε την άκρη του αεροδρομίου, τα πρώτα σπίτια της Φονταραμπή που είναι στα λίγα μέτρα και εκεί η πόλη του Αντάγη περίπου στα 700 μέτρα. Εδώ βλέπετε την άποψη του άξονα, ε, από τον άξονα ε, Ανατολής Δύσης, βλέπετε το κτίριο αυτό, 750 μέτρα από την άκρη της πίστας, εκεί είναι το νησί των πτηνών, όπως σας είπα, και το κτίριο αυτό θα στεγάζει τα γραφεία μιας ε, σημαντικής εταιρείας για την πόλη του Αντάχ. Όλοι γνωρίζουν τις οχλήσεις νομίζω, είναι παραδοσιακές οχλήσεις του αεροδρομίου, τριών τύπων μόλυνση, ηχητική, η οποία είναι τελείως ανυπόφορη. Οι συζητήσεις πρέπει να σταματούν στην Αντάι όταν προσγειώνονται τα αεροσκάφη η ατμοσφαιρική ρήπανση φυσικά, την, τα, γνωρίζετε το πρόβλημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και το πρόβλημα των υδρογονανθράπων γιατί η κυροζήνη ε, δημιουργεί πρόβλημα και τα υπολείμματα εναποτίθενται όχι μόνο στα σπίτια αλλά και σε ε, αλλού. Υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον. Η πόλη της ε, Διαρασόα ε, θεωρήθηκε Νατούρα το 2007, Νατούρα 2000, με συγχωρείτε. Η πόλη αυτή θεωρήθηκε ότι είναι ζήκο, είναι δηλαδή ε, ζώνη βιοπικιλότητας υγροτόπων και το έργο αυτό θα οδηγήσει σε καταπάτηση του κόλπου και της, ε, των συνθήκων για τα πτηνά. Αυτό, επίσης, η ύπαρξη των πτηνών δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Γι' αυτό ακριβώς θεωρείται επικίνδυνο το αεροδρόμιο και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι οι πιλότοι για να μπορούν να προσγειωθούν εκεί. Επίσης υπάρχει η υπερπτήση πάνω από τα κτίρια, υπάρχουν κτίρια πέντε ορόφων και βεβαίως ο κίνδυνος και πάλι είναι υπαρκτός. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί η Natura 2000 και ΖΙΚΟ, όπως επίσης και οι αεροπορικές αρχές έχουν θέσει το θέμα. Η επέκταση του διαδρόμου και η αύξηση του αριθμού των πτήσεων αποτελούν μια παράλογη κατάσταση. Θα πάρω το λόγο από τον συνάδελφο για ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Είμαι πρώην αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της, της Ακιτέν και σήμερα ασχολούμαι με την, περιοχή, με μεθόριο περιοχή. Ε, το θέμα των προδιαγραφών της ε, πίστας υπάρχει ένα κυνήγι κατά των, υπέρ των επιχειρήσεων εκεί. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Ναι, των ε, επιχειρήσεων ε, αεροπορικών εταιριών ε, χαμηλού κόστους και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα θέματα ανεργίας και οικονομικής κατάστασης. Ο οικονομικός κόσμος βεβαίως ασχολείται ελάχιστα με τους κατοίκους που είναι περίπου 100.000 η επέκταση αυτή παραβαίνει την, διακυβερνητική απόφαση διακυβερνητικής επιτροπής που υπογράφηκε στη Μαδρίτη το Μάρτιο του 1992 ώστε ε, το, αεροδρόμιο να μην ε, παραβιάζει ε, τις συνθήκες ζωής και ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής. Η σύμβαση αυτή περιόριζε σε 24 ημερησίω τις δραστηριότητες του αεροδρόμου. Αεροδρομίου σήμερα είναι γύρω στις 50 το καλοκαίρι. Επιπλέον, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιώδης λόγος η ευρύτερη περιοχή να έχει δύο αεροδρόμια που να απέχουν μεταξύ τους 33 χιλιόμετρα και κυρίως ε, να απογειώνονται μεγάλα αεροσκάφη για τουριστικούς προορισμούς. Θα είναι αρκετά απλό, αντίθετα, να υπάρξει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ του αεροδρομίου του Μπιαρίτς και της ε, ε, Φουενταραμπιά. Θα μπορεί ε, κανείς σε μισή ώρα από τη Φονταραμπία να βρίσκεται στο Πιαρίτ σε απολύτως λογική απόσταση. Αυτό γίνεται με την οργάνωση μιας μεταφοράς από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο και αυτό θα διευκολύνει τη ζωή και άλλων χρηστών και από τις δύο πλευρές της Μεθορίου η υφιστάμενη αρχή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για τη διαχείριση των αεροπορικών εγκαταστάσεων με τρόπο ε, καταμερισμένο και υπεύθυνο και όπως είπε ο συνάδελφος αυτό το έργο παραβαίνει τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου και άλλων αερίων θερμοκηπίου. Το διακύβευμα είναι να ξεκινήσει ένας ανταγωνισμός ε, και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτόν και να υπάρξει μια συμπληρωματικότητα από τις δύο πλευρές. Ε, γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ζητώ η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να είμαστε σε επιφυλακή για την, τους κινδύνους αυτού κατά των οικοσυστημάτων Natura 2000 και Ramsar για τους υγροτόπους τους, ε, σε περιοχές θαλάσσιες και ε, ποτάμις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ακούσουμε τον κύριο Σεβέρ Μαρτίν και πάλι εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Και πάλι το αντικείμενο της αναφοράς αυτής ε, αφορά ε, το δίκτυο Natura 2000 και μια περιοχή στην Ισπανία που ενδεχομένως μπορεί να προσβληθεί μετά από ε, επέκταση του αεροδρομίου της Ονταραμπία, ότι θα επηρεάσει τον κόλπο του Τσιγκούντι και την ίσο των πτηνών. Έχει οριστεί το Τζιγκούντι ε, ως ε, ζώνης ιδιαίτερης προστασίας των πτηνών ε, σύμφωνα με τις οδηγίες Habitat και την οδηγία για τα πτηνά. Σύμφωνα με την οδηγία του Habitat των οικοτόπων και το άρθρο 6.3 συγκεκριμένα, οποιοδήποτε έργο ή σχέδιο δεν συνδέεται άμετα, άμεσα συγγνώμη, με τη διαχείριση ενός ε, ε, τόπου Natura 2000 που μπορεί με τρόπο σημαντικό να επηρεάσει αυτούς τους τόπους θα πρέπει προηγουμένως να ε, υφίσταται μελέτη επιπτώσεων. Και μόνο εφόσον γίνει αυτή η έρευνα και αυτή η διαδικασία αξιολόγησης ε, τότε και μόνο τότε μπορούν να αποφανθούν οι αρχές με το, ε, για το έργο αυτό, γιατί δεν έχει σημαντική επίπτωση. σε ό,τι αφορά τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ε, πριν δώσουν την έγκριση για ένα έργο θα έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες. Πριν δηλαδή εγκριθεί η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα και βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχουν τροποποιηθεί στο μεταξύ ούτε διαψευστεί, ε, γνωρίζουμε ότι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου αυτού του έργου διεύρυνσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι καθοδόν γι' αυτό. Δεν έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες αρχές για το εάν ε, συνάδει, όχι συμμορφώνεται με τις οδηγίες. Δηλαδή δεν έχει δοθεί ακόμα σήμερα έγκριση. Άρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου και δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε παράβαση ή παραβίαση κοινωτικού δικαίου εφόσον δεν έχει εκδοθεί η παραβιαση κοινωνικού δικαιου Ευχαριστώ κυρία Όκεν. Ευχαριστώ και πάλι. Είναι ξεκάθαρο παράδειγμα αυτό. Θυμόσαστε την έρευνα που κάναμε στην Επιτροπή μας πέρυσι για το πόσο οι οδηγίες για την Natura 2000 αντιμετωπίζονται στα κράτη-μέλη. Ένα από αυτά τα οποία υπογραμμίσαμε με την έρευνα αυτή ήταν ότι όταν έχεις να χειριστείς ε, περιπτώσεις Natura 2000 πρέπει να βρεις ε, αποδεκτές εναλλακτικέ λύσεις. Ακούστε τι έχουμε εδώ. Έχουμε τρία αεροδρόμια σε μία μικρή ακτίνα. Κάτι άκουσα για 30 χιλιόμετρα περίπου. Είναι λίγο παράλογο να πηγαίνουμε προς την κατασκευή ενός μεγάλου αεροδρομίου σε μια τέτοια περιοχή. Υπάρχει εδώ το περιβάλλον, ο κόσμος, η ασφάλεια, η καθημερινή ζωή που όλα απειλούνται. Ε, λόγω αυτού του τεράστιου αεροδρομίου. Προσωπικά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αν θέλει κανείς να προσελκύσει τουρίστες, γιατί καταστρέφει τις ωραίες περιοχές. Καμιά φορά όμως αυτή η λογική δεν υφίσταται. Έχω δει τόσες και τόσες φορές, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά συχνά στην Ισπανία, αλλά όχι μόνο εκεί επαναλαμβάνω, ότι προσπαθεί κανείς να προσελκύσει όλους μπορεί καταστρέφοντας την περιοχή αλλά το θέμα είναι πρέπει να, ε, να δούμε μια ε, έρευνα, να, ζητήσουμε να γίνει μια μελέτη για εναλλακτικέ. Υπάρχουν εναλλακτικέ, εξ όσων γνωρίζω. Μπορούμε τώρα ήδη να απαντήσουμε ότι χρησιμοποιήστε τους πόρους και τη, τα ωραία τοπία σας με τρόπο περισσότερο προσεκτικό. Αυτά. sure, και να φροντίσουμε ότι η έρευνα να γίνει. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει. Ε, είναι τόσο σαφές, είναι τόσο προφανές. Είναι τόσο προφανές αυτό όλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουλάν. Πρόεδρε, γνωρίζω καλά αυτή την περιοχή, την νοτιοδυτική, πηγαίνω παλιά. Ήμουνα και διότι πιλότος ε, μικρό αεροπλάνο, ξέρω και το αεροδρόμιο. Και ξέρω τι είναι επαρκές το αεροδρόμιο. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συστήνει να γίνει μελέτη αντιχτύπου πριν το έργο. Είναι προαπαιτούμενο λογικό. Δεν ξέρω αν εμείς μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικέ. Η γαλλική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχομένω προτείνουν εναλλακτικέ, αν αποτύχει αυτό το έργο και το πρόγραμμα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετηθεί θετικά επί του προγράμματο θα αντέβαινε την υπεράσπιση, την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν θα ήταν κάτι λογικό. Από μια πρώτη ματιά θα έλεγα ότι αυτή η αναφορά είναι ευρέως αποδεκτή Πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τη μελέτη αντιχτύπου. Παρόλο που έχει ανασταλεί και έχει παγώσει το έργο, δεν μας εμποδίζει εμάς να τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά. εν αναμονή των εξελίξεων και βλεποντας κατά πόσο θα το έργο έχει. Ευχαριστώ. Ο κυριος Μπουστινάρο έχει το λόγο. Α, η κυρία Άουκεν παρεμβαίνει. Η κυρία Άουκεν διακόπτη. Έδινα το λόγο στον κύριο Μπουστινάρου και μετά εσείς. Ο Μπουστινάρου πρώτος. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι έχουμε εδώ. Έλλειψη ορθής εφαρμογής του Natura 2000 και της οδηγίας για τους βιοτόπους. Όταν μιλάμε για κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτοί πρέπει να εκτελούνται αυτομάτως. Τι ζητάμε. Να δούμε τα πορίσματα της αξιολογής περιβαλλοντικών συνεπειών. Κάτι που δεν έγινε ακόμα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Επιστολή στην τοπική αυτοδίκηση. Να υπενθυμεί στην τοπική αυτοδίκηση αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί κανόνε Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεύτερον, η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή έως ότου να λάβουμε μία απάντηση από τις αρχές και μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τελικά την όλη κατάσταση που σχετίζεται με το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ναι, κυρία Άουκεν. Είπα κάτι λάθος πριν. Ακτίνα 80 χιλιόμετρων, τρία αεροδρόμια. Και στα 30 χιλιόμετρα υπάρχει άλλο αεροδρόμιο. Από εμά εξαρτάται, θα έλεγα, να επιμείνουμε. Να βρούμε εναλλακτικέ. Έχουμε δικαίωμα και να πούμε και εμεί ότι και να μα λένε εκείνοι ότι υπάρχουν εναλλακτικέ. Γι' αυτό κάνουμε αποστολέ για να συλλέξουμε στοιχεία κλπ. και καμιά φορά επικροτούμε αποφάσει που παίρνουν οι αρχέ. Και εδώ είναι σαφέ ότι υπάρχουν εναλλακτικέ και αυτό είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό και για τους κανόνες των οδηγιών για την Natura 2000. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο ο αναφέρον. Πριν συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θέλω να πω ότι ένα ερώτημα σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και δεύτερον, όσον αφορά το φάκελο, υπάρχει μία απόφαση ε, τη, της ε, χωροταξικής έρευνας της νότιας χώρας των Βάσκων που είναι σαφής και ξεκάθαρη κατά της ε, κατασκευής ε, αυτής του αεροδρομίου. Ε, αναφέρει ότι επανειλημμένος ε, ε, επαναλαμβάνει ότι είναι κατά αυτής της κατασκευής. Σας ευχαριστώ. Μετά τις παρεμβάσεις του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικές σας, θεωρούμε ότι είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες που μας επέτρεψαν να το συζητήσουμε το θέμα. Αυτό που πρότεινε ο Χάρτης είναι αποδεκτό, αυτό που προτείνει και ο Μπαστονάρο. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών, πρώτα απ' όλα, καταρχάς. Υπάρχουν ανησυχίες πράγματι. Έχει γίνει μελέτη που δείχνει ότι εάν ε, χρησιμοποιηθεί γη πάνω από 5 εκτάρια, εάν επεκταθεί πολύ το έργο, θα υπάρχουν προβλήματα εξεπλάγινα από τις πληροφορίες που διάβασα εγώ στην έκθεση περιβαλλοντικών ε, συνεπειών. Άρα είναι σοφό να παραμείνει εκρεμές το θέμα ανοιχτή αναφορά αυτή, να δούμε τις εξελίξεις, να στείλουμε και μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές εκφράζοντας τις ε, ανησυχίες μας. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο και θα δώσω το, την Προεδρία ξανά στην Πρόεδρο μας. Πάμε λοιπόν στην αναφορά 23 που υπευλήθη από τον κύριο Γκέρχαρτ Χόλτσιγκερ και αφορά έναν αυτοκινητόδρομο στις ε, Καναρίους νήσους. Δεν είναι παρόν, παρόν αναφέρον. Δίνω το λόγο στον υπεύθυνο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας μιλήσει για το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η αναφορά 1400 του 2009 του κυρίου Χόλτσιγκερ όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αυτοκινητοδρόμου στις Καναρίες νήσους, στη Λαπάλμα. Εκεί ο αναφέρον καταρχάς ζητά να γίνει μια εκτίμηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του αυτοκινητοδρόμου που θα κατασκευαστεί μεταξύ Σάντα Κρούς Λαπάλμα και Λος Λιάνος Αριδάνε. Μετά εκφράζει την άποψη ότι οι ίδιοι στόχοι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μέσω διευρύνσεως δρόμων που ήδη υπάρχουν και θέτει τα θέματα κατά πόσο πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση από τα περιφερειακά ταμεία προς τις εξόχως απόκεντες περιοχές. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα προβεί σε κάποια σχόλια σχετικά με το ζήτημα. Όσον αφορά την χρήση των ε, περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης, εγώ θα έλεγα εκ μέρους της Γενικής Διευθύνσεως Ρίτζιο ότι οι Ισπανικές αρχές μας έστειλαν ε, πληροφορίες. Το πρόγραμμα αυτό του αυτοκινητόδρομου δεν δέχτηκε καμία χρηματοδότηση, δεν θα δεχτεί καμία χρηματοδότηση από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και περιφερειακών αρχών της ε, Ισπανίας. Το επόμενο που έχω να πω είναι ότι μοιράζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ανησυχίες του αναφέροντος δοθέντων των περιορισμών στη Λαπάλμα. Τα διευθυντικά ταμεία πράγματι θα πρέπει να εστιαστούν επί αναβαθμίσεως των ε, υπαρχουσών ε, υποδομών από το 2003 το 2006 στις Κανάριες νήσους τα λόγω ταμεία χρηματο, χρηματοδότησαν οδούς, αυτοκινητοδρόμους 40 χιλιόμετρα νέων ε, αυτοκινητοδρόμων και 130 χιλιόμετρα ε, έργων συντήρησης έλαβαν χώρα για τους υπάρχοντες δρόμους. Μοιραζόμαστε λοιπόν τις ε, ανησυχίες που εκφράζονται και αυτό είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται άλλωστε στα λειτουργικά μας προγράμματα. Όσον αφορά το 2007-2013 υπάρχει ε, θέμα προτεραιοτήτων που είναι η περιφερειακή και η τοπική δρόμη έχουν προτεραιότητα, οι περιφερειακοί δρόμοι, οι περιφερειακές οδοί μπορούν να βελτιωθούν για να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις με λιμένες και αερολιμένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί ένα τμήμα του σχεδίου για τις μεταφορές στα νησιά. Και αυτό ευθυγραμμίζεται και με τις επιθυμίες και τις ανησυχίες που εκφράζει ο αναφέρον. Ο συνάδελφος της Γενικής Διευθύνσεως ε, Περιβάλλοντος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βλέπουμε σε αυτή την αναφορά ότι αντιτίθεται σε ένα ε, έργο αυτοκινητοδρόμου στο Ινίσο Λαπάλμα, στα Κανάρια νησιά. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται να συμπληρώσει τα όσα είπε συνάδελφος από την περιφερειακή πολιτική. Όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, σε αυτό το αυτοκινητόδρομο εφαρμόζεται πλήρως η Οδηγία 85337 για τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, διαφόρων έργων ε, ιδιωτικού και δημοσίου με σύμπραξη. Υπάρχει το παράρτημα 1 που αφορά έργα τα οποία αποχρεωτικά πρέπει να είναι αντικείμενο περιβαλλοντικής μελέτης και το παράρτημα 2 η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και ε, ταχαίων οδών είναι ε, στο παράρτημα 1 και μάλιστα ε, στο εδάφιο 7β. Και χρειάζεται βεβαίως πάντα πρώτερη μελέτη. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, σημαίνει περιγραφή καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων πριν δώσει την έγκριση ενδεχομένω η αρμόδια αρχή. Το κοινό μπορεί να εκφράσει την άποψή του, ε, γίνονται διαβουλεύσεις με μία σειρά από αρχές και το αποτέλεσμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν δοθεί η άδεια. Και θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται το κοινό για το περιεχόμενο της έγκρισης θα πρέπει να πούμε ότι με βάση την πληροφόρηση που έχουμε είναι πάρα πολύ πρώιμο ακόμα το στάδιο του έργου και θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει τις παρατηρήσεις του επιτόπου αφού είναι στο στάδιο ακόμα που γίνεται η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Είναι Πρόημο αυτή τη στιγμή να πούμε εάν ε, έχουμε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επέμβει περισσότερο σε αυτό το θέμα, αφού όπως είδαμε αφενός δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου και επιπλέον βρίσκεται σε ε, πάρα πολύ πρώιμο στάδιο, είπαμε, και δεν μπορεί ακόμα να αποφανθεί κανείς, γιατί δεν έχει γίνει καν η μελέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος Μπουστενάρο έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, μόλις μας ενημέρωσε η Κομισιόν ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε αυτό το έργο, αλλά η, ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ε, υποχρεωτική, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να περιμένουμε τη στιγμή που θα γίνει η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο οι ανησυχίες του αναφέροντος αλλά και άλλων εμπλεκομένων θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα και πώς αυτή η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επισημάνει τα προβλήματα ε, στο περιβάλλον. Να μείνει ανοιχτή λοιπόν μέχρι τότε. Αυτό προτείνω. Okay. Λοιπόν, κοινή προσέγγιση να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά εν αναμονή εξελίξεων. Περνάμε στις δύο αναφορές του σημείου 24 του σημείου 24 λοιπόν αναφορά 764 και 133 του Φιλίπ Ρικλέ και του Ζων Ανουί Ντιβάλ δεν είναι παρόντες οι αναφέροντες και σε αυτή την περίπτωση θα δώσω το λόγο στον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γκριμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με σκοπό να σας παρουσιάσω την κατάσταση σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των δύο αναφορών, θα σας αναφέρω σε τέσσερα σημεία ε, το αντικείμενο αυτών των αναφορών και περί τίνος πρόκειται. Τα επιχειρήματα του αναφέροντος, τις δράσεις της Κομισιόν σε σχέση με το περιβάλλον για την αντιμετώπιση αυτών και το γεγονός ότι αυτό ε, είναι αντικείμενο ε, δίκης που έγινε σε Διοικητικό Δικαστήριο της Γαλλίας, το οποίο απεφάνθη και τέλος την τεχνική και νομική ανάλυση που έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος υπό το φως των πληροφοριών που ε, λάβαμε. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ένα έργο ψυχαγωγίας ε, και διακοπών, ένα πάρκο ψυχαγωγίας και διακοπών, που θα αποτελείται από, 150 περίπου ε, κατοικίες, μια ανοιχτή πισίνα, δύο χώρους στάθμευσης, ένα χώρο υποδοχής και ένα αστικό δίκτυο που θα χειρίζεται όλα αυτά τα έργα υποδομής. Στόπος είναι, είναι λοιπόν μια, είναι μια μεγάλη τουριστική επιχείρηση της Γαλλίας η οποία ασχολείται με αυτό. Θα γίνει αυτό στο, στην περιοχή Duizon, Loire σε μια ε, περιοχή που η Γαλλία έχει ε, εντάξει στο ε, δίκτυο Natura. Υπάρχει ιδιαίτερη ε, προστασία των πτηνών που η Γαλλία την έχει εντάξει στην οδηγία προστασίας των πτηνών. Έγινε λοιπόν μια διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για να διαπιστώσουμε αν το σχέδιο κάλυψης του ε, άλλαξε και δόθηκε στον ανάδοχο το 2007 μία άδεια οικοδόμησης μαζί με άλλες δύο τροποποιητικές άδειες οι οποίες χορηγήθηκαν το 2008 και η τελευταία το Μάρτιο του 2010. Ε, Γιατί αυτές οι τροποποιητικές άδειες, επειδή οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, η η ε, γνωμοδότησε υπέρ υπό επιφυλάξεις. Έτσι λοιπόν, ε, για να καλυφθούν οι επιφυλάξεις, έγινε αυτή η τροποποίηση της άδεια οικοδόμησης. Ποια είναι τα επιχειρήματα των αναφερόντων. Είναι κυρίως τέσσερα. Πρώτον, υποστηρίζουν ότι το έργο αυτό δεν θα έπρεπε να έχει αδειοδοτηθεί δεδομένου ότι θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή που είναι Natura 2000. Επίσης, δόθηκε άδεια χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έπρεπε να έχει γίνει εκ των προτέρων. Η Natura 2000, ε, μελέτη για την Natura 2000 είναι ανεπαρκής όσον αφορά τις επιπτώσεις του έργου και τέταρτον το έργο αυτό θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στους δύο ε, λίμνες, ε, στις δύο δεξαμενές γύρω από τις οποίες θα κατασκευαστεί. η Κομισιόν και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ασχολήθηκε. Καταρχήν ανοίξαμε μια διαδικασία παράβαση κατά της Γαλλίας το 2008. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έστειλε δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσε πληροφορίες από τη Γαλλία. Στην αρχή δεν λάβαμε απάντηση. Ξεκίνησε διαδικασία παράβασης για μη συνεργασία. Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 2008. Κατόπιν ε, εστάλει Επιτροπή ε, Επιστολή όχληση προς τη Γαλλία, κατά την οποία οι γαλλικές, μετά την οποία οι γαλλικές αρχέ έδωσαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η διαδικασία λοιπόν αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010 μετά από την αποστολή των πληροφοριών και των στοιχείων που είχαμε ζητήσει από τις αρχές. Πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα υπήρχαν επιστολές ε, που ζητούσαμε πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές, τρεις μάλιστα, ζητώντας ε, διευκρινήσεις, ε, πληροφορίες, ε, τεκμηριώσεις. Υπήρχε μια αρκετά ογκώδης ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κομισιόν και των Γαλλικών Αρχών. Απήντησαν πέντε φορές οι Γαλλικές Αρχές και έχουμε στείλει σημαντικό όγκο ε, εγγράφων, Natura 2000, τα σχέδια του ε, έργου κτλ. κτλ. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν να γίνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου αυτού. Το τρίτο σημείο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι το εξής. Το έργο αυτό το ε, χειρίστηκε το Διοικητικό Δικαστήριο της Γαλλίας στην Ορλεάνη. Η Ένωση για την προστασία της περιοχής προσέφυγε στο δικαστήριο για να ζητήσει την ακύρωση της άδειας οικοδομής που χορηγήθηκε στο έργο. Στις 16 Ιουνίου του 2009 ο διοικητικός δικαστής είπε ότι αρκούσε το Natura 2000 και ότι ήταν πλήρης η αίτηση για την αδειοδότηση και δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το έργο αυτό θα επηρέαζε σημαντικά την περιοχή αυτή και γι' αυτό αθωώθηκε. Κατόπιν έγινε η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο της Νάντης ζητώντα την ανέρεση της προηγούμενης απόφασης. Σήμερα μάθαμε ότι το δικαστήριο της Νάντης θα ε, δικάσει στις 25 Μαρτίου του 2011 την υπόθεση αυτή και η απόφαση θα ε, ληφθεί τον Απρίλιο. Θέλω απλώς να αναφέρω στο γεγονός ότι υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2009 για τις συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών όπου αναφέρεται ότι στο σημείο ΚΑΠΑ ότι υπάρχει μια διαδικασία μεταβίβασης των, ε, ε, και υπάρχει θέμα διαδικασίας ενώπιον των εθνικών αρχών για την επανεξέταση των αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, ο Γάλλος διοικητικός δικαστής έχει αρμοδιότητα και υποχρέωση να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο, να εφαρμόσει, να ερμηνεύσει το εθνικό δίκαιο υπό το φως του κοινοτικού δικαίου. Φυσικά λοιπόν τα εθνικά δικαστήρια είναι η πρώτη θέματοφύλακες της καλής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου παρά το γεγονός ότι ο δικηγός δικαστής της Γαλλίας ε, δήλωσε ότι η άδεια είναι ε, ισχυρή, οι, επιτροπές, η Επιτροπή μελέτησε τεχνικά το θέμα, χωρίς να ξέρουμε ότι είχε φτάσει υπόθεση στο διοικητικό δικαστήριο. Αναλύσαμε λοιπόν τα συμπεράσματα της Κομισιόν, υπό το φως των πληροφοριών που είχαμε, είναι ότι δεν υπάρχει εμφανής παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και κάτι το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε σε σχέση με αυτό το έργο. Καταρχήν, ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι ε, δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί άδεια λόγω του χώρου. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η οδηγία για τους οικοτόπους δεν μπορεί να απαγορεύσει οποιοδήποτε έργο επειδή θα επηρεάσει κάποιο χώρο. Υπάρχει ένας, μια ρήτρα που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προστατεύουν τους χώρους και τα είδη στο, στο βαθμό που δεν θα είναι σημαντικές οι επιπτώσεις, δηλαδή ε, δεν θα υπάρχει έργο που θα θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον ή ε, την, ε, τις συνθήκες διατήρησης ενός είδους υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά αν οι επιπτώσεις αυτές δεν θεωρούνται σημαντικές, τότε η οδηγία για τους οικοτόπους δεν έχει υποχρέωση να απαγορεύει. Και το 3.6 και το 3.7 αναφέρεται στο τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις των, ε, ε της Natura 2000. Το έργο από ό,τι μάθαμε, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το χώρο αυτό, την περιοχή Σολόνια. Έγιναν δύο μελέτες Natura 2000 με συμπέρασμα που συμπίπτει με τις ε, περιβαλλοντικές αρχές περιοχής που κατέληξαν ότι η τα μέτρα του έργου ε, μπορούν να προστατεύσουν την περιοχή. Μόνο, μία, σε μία περίπτωση θα υπήρχε επίπτωση σε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν θεωρείται προτεραιότητος στην, από τη διαδικασία των οικοτόπων. Και αναφέρει ότι η, αναφέρεται ότι η ακύρωση της άδειας ε, οικοδομής ε, πρέπει να γίνει μόνο σε περίπτωση που θα υπάρχει έμεση ή άμεση επίπτωση στην περιοχή. Επίσης, το έργο δεν θα έχει επίπτωση, σημαντική επίπτωση στην ζώνη ειδικής προστασίας που αφορά τα πτηνά και η οποία βρίσκεται σε κάποια απόσταση από εκεί, τη ZPE. και η οποία ζώνη έχει καθοριστεί για την προστασία ενός συγκεκριμένου είδους. Αυτά ε, αποφασίστηκαν το 2009. Δεύτερο επιχείρημα του αναφέροντος δόθηκε η άδεια χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπό την έννοια της ε, οδηγίας του 96. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτού του είδους τα έργα αναφέρονται στο παράρτημα 2 της οδηγίας, όπου υπάρχει κατάλογος έργων για τα οποία η αρμόδια αρχή είναι αυτή που αποφασίζει εάν υπάρχει υποχρέωση ε, για εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που μας ε, κάνουν να θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο εδώ. Έχουμε κάνει, υπάρχουν δύο μελέτες Natura 2000, μία μελέτη για τους υδάτινους πόρους κλπ. Τρίτον, οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι είναι ανεπαρκείς οι μελέτες Natura 2000, δεν έγιναν την κατάλληλη στιγμή και δεν μελετήθηκαν αυτά που έπρεπε να μελετηθούν. Εδώ έχουμε δύο μελέτες Natura 2000. Η μία έγινε το 2005 και η DIREN, η αρμόδια αρχή, ε, γνωμοδότησε κατά λέγοντας ότι δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη εποχή αυτή η μελέτη. Η Natura 2000 ε, ακριβώς ε, Έγινε, επανελήφθη λοιπόν η μελέτη αυτή του Natura 2000 γιατί προ, για την πρώτη ίσχυαν αυτά τα οποία λένε οι αναφέροντες. Το συμπέρασμα της περιφερειακής αρχής, της αρμόδιας ε, περιφερειακής αρχής είναι ότι το, ο φάκελος του Natura 2000 περιλαμβάνει μια σειρά από που μας επιτρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένα τις επιπτώσεις. Τέλος, οι αναφέροντες αναφέρονται για τις δύο δεξαμε, στις δύο δεξαμενές ε, υδάτων που υπάρχουν. Και βεβαίως αυτές είναι σημαντικές για την καλή λειτουργία του οικοσυστήματος της περιοχής. Πρόκειται για ένα θέμα ε, υδάτων της βροχής. Πώς θα συγκεντρώνονται αυτά αρχικά προβλεπόταν να μπαίνει στις δεξαμενές κατευθείαν αυτό το νερό της βροχής, κατόπιν μετά από αρνητική γνωμοδότηση επανεξετάστηκαν τα σχέδια του έργου και χρησιμοποιήθηκε η άλλη εναλλακτική για την οποία δόθηκε ε, το πράσινο φως από την αρμόδια αρχή. Αυτά κυρία Πρόεδρε έχω να πω για τις δύο αυτές αναφορές. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Άουκεν. Εν συντομία, ξέρετε αν ο αναφέρον ζήτησε γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως μπορεί να γίνει έχουν τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όχι δεν υπάρχει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ο αναφέρον μισό λεπτό λέει η Πρόεδρος να μαζέψουμε και τις ερωτήσεις, να ακούσουμε και την άλλη ερώτηση. Ο κ. Βαλά. Ναι, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι ερώτημα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαβήματα, διακόπτει ο μιλητής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ φανταζόμουν ότι ήθελα να ακουστεί άλλη μια ερώτηση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τελικά σε αυτά που ρώτησε η συνάδελφος Άουκεν. Εκτός μικροφώνου Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πήγαν στο διοικητικό εφετείο της ΝΑΝΤ. Θα τοποθετηθεί το δικαστήριο, θα γνωμοτήσει τέλος Απριλίου, Απρίλιο-Μάιο του 2011, ανάλογα με την απόφαση. Αν αναφόρον κάνει έφεση, θα πρέπει να πάει στο, νότο, το, στο Συμβούλιο Επικρατείας αν έχει αντίρρηση όσον αφορά την τοποθέτηση του δικαστηρίου της ΝΑΤ. Ο συνάδελφος Μπολάου έχει το λόγο. Ναι, νομίζω ότι όλες, όλα τα διαβήματα έγιναν σύμφωνα το γαλλικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο στη γαλλική επικράτεια μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν αυτή η αναφορά ως ε, κλεισμένη, μπορεί να κλείσουμε την αναφορά. Καλώς λέει. Υπάρχει γενική συμφωνία να κλείσει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάω στην τελευταία αναφορά του κυρίου Νταν Μπρέναν που αφορά μια εικαζόμενη μόλυνση κάποιων εκμεταλλεύσεων κτηνοτροφικών. Όσον αφορά αυτήν την αναφορά, έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωμα από τις πλευράς της Ormond Brick που απαντά σε αυτά που αναφέρονται στην ε, αναφορά. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα για να κάνει την παρέμβασή του. Λοιπόν, ευχαριστώ την Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ την Επιτροπή που με κάλεσε σήμερα να παρουσιάσω το θέμα. Είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζω ε, το θέμα. Ε, τα προβλήματα στο αγρόκτημά μου είναι πολύ σοβαρά και οφείλονται σε σοβαρή περιβαλλοντική βλάβη. Το εργοστάσιο σταμάτησε την παραγωγή του το Δεκέμβριο του 2008. Από τότε έχει αυξηθεί η ανάπτυξη των, ε, σε σχέση με την, περίπτωση, με την περίοδο που ήταν ανοιχτή που ήταν ανοιχτό το εργοστάσιο. Χρειαζόμαστε διαβεβαίωση ότι θα, θα ασκηθεί πίεση στι Ιρλανδικέ αρχέ για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα επιτραπεί να ξανασυμβεί. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα, θα γίνει η πίεση στις Ιρλανδικές αρχές για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν θέλω να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν ξέρω τι επιπτώσει έχει αφήσει αυτό το αγρόκτημά μου. Ήρθα εδώ ε, ε, μαζί με μια ομάδα ε, επιστημόνων, στους οποίους θα ήθελα να, επιβάλλετε ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Τόμ Σέβεν και είμαι ερευνητής σε Είμαι κτηνίατρος. σε μεγάλα ζώα. Ήμουν, ε, ε, τα τελευταία 6 χρόνια εργάζομαι στην εκτροφή του. Τον Ιανουάριο το 2003 οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας άρχισαν έρευνα για, το, για λόγο που μειώθηκε σοβαρά η παραγωγή. 18 μήνες μετά εξέδωσαν προσωρινή έκθεση που έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία νόσος. Και απέκλεισε τη σαλμονέλα η χρόνια πνευμονία. Και ότι έλεγε ότι τα ζώα ήταν εντάξει. Επίσης, αυτό επαναλήφθη το Μάιο του 2005 δεν είχαν βρει καμία ασθένεια που να είναι υποκείμενη του προβλήματος. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, οι περισσότερες ε, ασθένειες που ε, βρέθηκαν στην Ιρλανδία θεωρήθηκαν ε, εν μέρη υπεύθυνε για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και οι υποτιθέμενες ασθένειες ξαφνικά εμφανίστηκαν όταν ε, βγήκε η έκθεση. Μετά το 2007 ε, πάλι δηλώναν ότι δεν υπήρχε ένδειξη σημαντικής νόσου. Το 2005 ε, σφαγιάστηκαν ε, μερικά νεαρά ζώα και έγινε και νεκροψία και μετά από τέσσερις μήνες, πέρα από κάποιες μικρές πνευμονοπάθειες, είχαν προβλήματα στο λεπτό έντερο. Επίσης, ε, στο σκελετικό σύστημα. Ε, ο χόνδρος είχε παραμείνει ε, λεπτός και δεν είχε γίνει οστό. Οι ορμόνες αυξητικές δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να ήταν. Και οι μαλακίστοι, όπως η καρδιά και ο πνεύμονας, είχαν διηθηθεί από στέινη μάζα. Δηλαδή το κόκαλο πήγαινε και στα μαλακά μόρια αντί να γίνει κόκαλο, εκεί που έπρεπε και από πλευρά ε, ανθρώπινη υγείας θα έπρεπε να ε, αρχίσουν να χτυπούν διάφορα ε, καμπανάκια, αλλά θεωρήθηκαν αμεληταία αυτά τα ευρήματα και αυτό αφορά διάφορους ιστούς που έχουν να κάνουν με προβλήματα οστεοπόρωσης και μαλακά οστά. Λοιπόν, δεν εντοπίστηκαν σωστά, δεν απομονώθηκαν τα άρρωστα ζώα Η Σεβίρα ήταν το, ο όμιλος που έκανε αυτή την έρευνα, ε, αλλά ήταν κατακαιρματισμένη η έρευνα μόνο μερίς. Ε, αν ήξερε ότι είχαν πρόβλημα τα ζώα του, ο εκτροφέας θα τα είχε απομονώσει και δεν θα τα έστρεψε στην αγορά. Έκλεισε το εργοστάσιο και όταν σταμάτησε η παραγωγή, Αυξήθηκε η γαλακτοπαραγωγή ημερήσια ε, από 2,1 κιλά την ημέρα από 0,21 σε 0,78 την ημέρα. Αναζώ. Ε, υπερ, διπλασιάστηκε. Ήταν πολύ χαμηλά τα επίπεδα ε, σελινίου αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Ε, ακόμα και αν τους έδιναν. Ε, όταν υπάρχει κάδμιο στα κύτταρα, ε, είναι καλύτερο να παίρνεις κάδμιο και να αφήνεις το σελήνιο ως δείκτη. Αυτό τι σημαίνει όταν προσλαμβάνουν τα κύτταρα, βαρέα μέταλλα, κάδμιο, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να διατηρήσουν ε, τη δραστηριότητά τους και δεν ε, διατηρούν τα μέταλλα που χρειάζονται και εμφανίζουν μεγάλες ανεπάρκειες. Είναι άμεσες και έμεσες τοξίνες και ε, αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις ανετικές σε ζώα στην ανάπτυξή τους, νεαρά. Και ιδιαίτερα η έκθεση σε ραδιενέργεια ε, επηρεάζει πάρα πολύ το ε, τοξίκωση τελικά από κάδμιο ε, αυξάνει τις μεταβολικές νόσους και τις ορμονικές νόσους. Και αυτό διαπιστώθηκε από το 1992 στην εκτροφή αυτή. θα μπορούσα να προσθέσω ότι για το 2006 και 2009 οι εκθέσεις που εξεδόθηκαν ε, ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητικές και φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ιρλανδία. Και ξέρω ότι έχουν γίνει αντίστοιχε και σε πανεπιστήμιο. Members. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι ο Σάιμον Χάιτ, είμαι περιβαλλοντολόγος, χωρίς μικρόφωνο, Α. και εκπροσωπώ την ε, Ιρλανδική Ένωση Αγροτών. Είμαι καθηγητής στο Λίμερικ και έχω ασχοληθεί ερευνητικά με τη χημεία. Δεν εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο ενώπιν της Επιτροπής σας. Μου γνωστοποίησαν την περιοχή, την, το πρόβλημα ε, το 2005 το 2000, τον Ιούλιο του 2007 η σημασία της περιβαλλοντικής βλάβης στην εκτροφή ήταν σαφής για τα μέλη που επισκέφθηκαν την εκτροφή. Πέρυσι, μετά ε, τη δημοσίευση της έκθεσης Σιβερίεν ήρθαμε στην Επιτροπή για να υποβάλουμε τους λόγους της ανησυχίας μας ε, ότι δηλαδή δεν έλεγαν την αλήθεια για την υπόθεση αυτή. Έκτοτε είδαμε μία προσθήκη στην, ε, στην έκθεση Σεβίρ και μία προσθήκη στην έκθεση που αφορούσε την έρευνα. Έγινε μια έρευνα το 2006, η οποία εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ήταν τόσο εσφαλμένη, που θεωρήσαμε ότι το Υπουργείο θα ντρεπόταν να την δείξει και όχι να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την αλήθεια. Στο διάστημα αυτό έγιναν περιβαλλοντικές μελέτες στην εκτροφή γιατί διαπιστώθηκε ότι η ζωή των φυτών, κυρίως τα δέντρα και η θάμνη, κατά καιρού ε, ε, υπέστησαν σοβαρή ζημιά. Επίσης η επιρροή, η ζημιά αυτή ε, οφειλόταν σε ε, ε, ατμοσφαιρική μόλυνση. Ήταν περιορισμένη σε μια περιοχή του, της εκτροφής και όχι στον περιβάλλοντα χώρο. Η, περνούσε μέσα από τα φύλλα η μόλυνση και πολλές φορές τα κατέστρεφε. Υπήρξε και νέα ζημιά και κακή υγεία στα ζώα της εκτροφής. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη συσχέση τα συμβάντα αυτά ήταν, συνέβαιναν μόνο όταν λειτουργούσε το ε, εργοστάσιο παραγωγής πλήνθων και όχι όταν σταματούσε. Οι χημικές ουσίες του ε, που έπεφταν στο νερό κατά πάσα πιθανότητα ήταν ε, αυτές που προκαλούσαν τη ζημιά. Διάφορες, διάφορα φθοροπαράγωγα. Έχουμε εκθέσεις φορέων και διάφορες εξηγήσεις οι οποίες πραγματικά είναι απίστευτες τα, οι ενώσεις του φθορίου αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ε, αναφερόντουσαν μόνο κατά το ίμιση γιατί ε, δεν ήταν σωστές οι μετρήσεις των ε, συσκευών. Οι υπολογισμοί λοιπόν στηριζόντουσαν σε εσφαλμένα στοιχεία. Η έρευνα που έγινε από το EPA έκανε μία μελέτη υγείας των ε, ζώων και των ε, δένδρων. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν τελείως απαράδεκτο. Τα ευρώματα λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με την ε, εκτροφή. Η μελέτη της υγείας των δένδρων αναφέρθηκε και στη μόλυνση και στη ζημιά, αλλά ανέφερε ότι η μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι ρήποι που είχαν προκαλέσει τη ζημιά και αναφέρθηκε και ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά κάποια επίπεδα φθορίου. Όταν όμως αναλύθηκαν τα δείγματα, η ανάλυση έγινε μήνες μετά από τη στιγμή που φάνηκε ότι είχαν επηρεαστεί τα ε, φυτά. Δεν εντοπίστηκαν τα, ε, οι ουσίες στα φυτά που σημαίνει ότι δεν καταστράφηκαν από αυτές δεν είναι σωστός τρόπος γιατί αυτές είναι εξαιρετικά πτυτικές ουσίες. Οι εκπομπές όπως φαίνεται στην έκθεση Σεβίρ μοιάζει ότι ε, τα φυτά επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις ημερήσιες και οριές συγκεντρώσεις των ουσιών. Και πάλι η έκθεση δείχνει ότι οι πολύ ψηλές συγκεντρώσεις του καδμίου συγκεντρώνονται σε κάποιο σημείο της εκτροφής. Επισημαίνεται ε, διοξίδιο του θείου, βαρέα μέταλλα και πτυτικά ε, και αέρια εκπομπών. Υπάρχουν πάρα πολλές, ε, πολλά στοιχεία όλων των εκθέσεων που δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα οι ρήποι που προκαλούν αυτή τη, ζημί, τη ζημιά προέρχονται από το εργοστάσιο πλήνθων που παράγει τους ρήπους αυτούς. Και επίσης δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι η ίδια ε, ε, ρήπανση που κατέστρεφε το νερό και τη, τα φυτά θα, θα δημιουργούσε προβλήματα και στα ζώα. Ο συνδυασμό των παρένων μετάλλων με τι άλλε αυτέ χημικέ ουσίε σαφώ εξηγεί τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στα ε, βοηδή, όπω με ενημερώνουν και η κτηνίατρη. Το 2010 μια περαιτέρω περιβαλλοντική μελέτη που έγινε έδειξε ότι δεν υπήρχε περαιτέρω σημειά στα φυτά από το 2008. Μέχρι τον Ιούλιο του 2010 η αναγέννηση των φυτών και των δένδρων της περιοχής ήταν σημαντική. Ακόμα και τα φυτά που μοιάζαν τελείως νεκρά το 2008 είχαν ανακάμψει. Η πυκνότητα των ε, δένδρων ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό συμπίπτει με τις δικές μου παρατηρήσεις στα ζώα της εκτροφής που βελτιώθηκε η κατάστασή τους κατά πολύ. Και αυτό στηρίζεται και από την ε, βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής. Όλες αυτές ε, οι αλλαγές συμπέπτουν με, την, με τη διακοπή της λειτουργίας και τη σταμάτημα των ρήπων. Εγώ θεωρώ ότι οι έρευνες που προσπαθούν να βρουν ε, τα αίτια για κάθε κομμάτι είναι ασήμαντες. όπως τα κομμάτια ενός puzzle, η σημασία κάθε κομματιού είναι εμφανής όταν αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Όταν δει κανεί τη συνολική εικόνα μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μπορείτε να φανταστείτε τι εκνευρισμό αισθάνεται κανείς όταν ε, κανείς αισθάνεται ότι τα προβλήματά του αντιμετωπίζονται από ανθρώπους και δεν δημιουργούν μια συνολική εικόνα ε, για, να είναι, ε, για να μην δυσαρεστηθούν κάποιοι. Κάνω έκκληση. Σας παρακαλώ να δεχτείτε ότι αυτή η αγροτική οικογένεια έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, έχει αποστεί ζημιές και άγχος από τέτοιες απώλειες. Αλλά επίσης ε, αυτές οι ε, η προσβολή κατά της αξιοπρέπειάς του με όλα αυτά που έχουν υποθεί είναι μεγάλη και είναι σημαντικό αυτό και για πολλούς άλλους οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωση. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον δόκτωρα J.J. Λίχη. Um, Νομίζω για να ξεκινήσει η συζήτηση δεν θα έπρεπε να πούμε πολλά περισσότερα για την ώρα. Καλώς. Στον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσω το λόγο τώρα. Thank you, Madam President, and... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχολιάσει ξανά στο παρελθόν την αναφορά αυτή. Και έκτοτε έχουμε προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναλύωτα τα συμπεράσματα. Ε, εξετάσαμε αυτό το θέμα του πληθοποιού με την Ιρλανδία και τα επιχειρήματα ε, του ε, αναφέροντος και τα επιχειρήματα των Ιρλανδικών αρχών. Μας έδωσαν κάποιες ε, πληροφορίες που γέννησαν και νέα ερωτηματικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προς την Ιρλανδική κυβέρνηση, ειδικά σε σχέση με την άδεια για την εγκατάσταση αυτού του εργοστασίου, τον τρόπο λειτουργίας και τι ε, αποτελέσματα έδωσαν οι επιθεωρήσεις των αρμοδίων Ιρλανδικών αρχών. Δώσαμε ιδιαίτερα προσοχή στη ρήπαση με κάδμιο και το λειτουργικό καθεστώς ε, του ίδιου του εργοστασίου. Όπως είπε και ο ε, αναφέρον από την αρχή, έχει σταματήσει τώρα η λειτουργία της εγκατάστασης, έχει κλείσει ε, το πληθοποιείο, αλλά οι πληροφορίες μας έχουν δοθεί όταν λειτουργούσε ακόμα. Ιδιαίτερα η άδεια λειτουργίας που δόθηκε από τις αρμόδιες αρχές ε, ε, στα πλαίσια της σας οδηγίας. Μελετήσαμε και τις οριακές τιμές για την ρήπανση, τις επιτρεπόμενες ενώ. και αυτές ήταν ε, σύμφωνες ε, με την οδηγία IPPC. Ζήτησαμε και νέα πληροφόρηση από τις Ελλαδικές Αρχές για μελέτες που έγιναν για το θέμα αυτό έκτοτε και όπως αναφέρεται και στην ενημέρωση που πήραμε, επιβεβαιώθηκε η ρήπανση με κάδμιο σε επίπεδα που μπορούσαν να οδηγήσουν μεν στα όσα λέει ο αναφέρον, αλλά οι μελέτες δεν ε, το απέδειξαν αυτό. Τι γίνεται με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά ε, βάσει του υλικού που μας έστειλαν και την ε, άδεια για το IPPC, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου, εμείς δεν ε, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πούν κάτι. Ε, Μακίνες. Κυρία Μακίνες, δεν ζήτησα το λόγο τώρα, σε λίγο θα ζητήσω το λόγο. Δεν σήκωσα το χέρι μου ακόμα, δεν σήκωσα το λόγο. Ο Γενικός Γραμματεύς μου είπε ότι στήσα το λόγο. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Γιάρα. Äh, Αυτό είναι μια ερώτηση προς τους αναφέροντες, γιατί έχουμε τώρα το πρόβλημα, προφανώς. Έχει μεγάλες ζημίες υποστεί η εκτροφή Άλλωστε αυτό είναι αποδεδειγμένο και απειλούν την ίδια την επιβίωση και τη λειτουργία της ε, τροφής. Αιτία υπάρχει, πολύ ψηλή μάλλον περιεκτικότητα σε κάδμιο, υποτιθέμενη όμως, η καζόμενη όπως λέω. Απόθεν αυτό το, το κάδμιο, ο αναφέρον λέει ότι είναι το εργοστάσιο το, δίπλα το πληθοποιείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν έχουμε αποδείξει αυτό, δεν υπάρχουν αποδείξεις γιατί όλες αυτές οι τιμές που ελέγχθησαν ήταν ε, επιτρεπτές, υπήρξε κάποια απόκληση, αλλά έφτιαχε λέει το μηχάνημα Μέτρηση. το όργανο. Εγώ θα το πω δηλητηρίωση από κάδμιο, ναι, ήταν τοξική, ε, αλλά μπορούμε να αποδείξουμε ότι προέρχεται από το εργοστάσιο αυτό παραγωγής πλήθων. Υπάρχει μια ένδειξη όμως, από τότε που έκλεισε, που σταμάτησε τη λειτουργία της, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα φαινόμενο που μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Α, κατά τα άλλα πρέπει να πω επίσης ότι οι αξιώσεις για τις αποζημιώσεις θα πρέπει να τεθούν σε εθνικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ναι, Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν κάνω την παρέμβασή μου. Αυτό το πλυνθοπείο προσεκλήθη στην συνάντηση. Παρίσταται εκπρόσωπος του πλυνθοπείου εδώ. Έγραψαν ένα σημείωμα το οποίο είναι στο φάκελο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγγνώμη, ζήτησα κάτι άλλο. Τους καλέσατε. Είναι παρόντες. Υπάρχει εκπρόσωπος εδώ. Πάντα καλούμε εκείνους που είναι διαθέσιμοι. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος αυτής της εταιρεία. Να, να, να, να τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω τους αναφέροντες και τους εμπειρογνώμονες την ομάδα αυτή και ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα την αρχή του θέματος. Ατυχώς ήμουνα σε άλλη συνεδρίαση. Όπως ο συνάδελφος Πίτερ Γιάρ είπε, υπάρχουν και καλά μαντάτα. Βελτιώθηκε η κατάσταση στην εκμετάλλευση. Το πρόβλημα όμως για την οικογένεια του Νταν Μπρέναν και τον Νταν Μπρέναν είναι ότι δεν ε, λύσαμε πλήρως, δεν τα αίτια. Επί σειρά ετών συνέβαινε αυτό. Άκουσα, διάβασα την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή τεχνική. Λέει ότι είδαμε τα στοιχεία που μας έδωσαν οι αρμόδιες αρχές και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διάβασα και την επιστολή από το πληθοπείο που είναι αρκετά λεπτομερής. Ανέφερε τη δική τους θέση σχετικά με αυτά που ακούσαμε στην αναφορά. Θεωρώ ότι έχουμε αποτελματωθεί, έχουμε βαλτώσει. Ο Νταν Μπρέναν δεν είναι ικανοποιημένο, δεν θα έχει ικανοποίηση έχει κολλήσει σε αυτές τις δυσκολίες επί πολλά χρόνια και εγώ δεν μπορώ να δω εμείς σαν Επιτροπή Αναφορών πώς να βοηθήσουμε. Άκουσα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άκουσα αυτά που είπε και ο Πίτερ Γιάρ ε, που είπε για την αποζημίωση, ότι πρέπει να, γίνει, να δοθεί αποζημίωση σε επίπεδο κράτους μέλους. Άρα έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα μπροστά μας. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ο, σύμφωνα με τα οποία α, προβληματίζονται και τα δύο μέρη και δεν υπάρχει επιστημονική επιτροπή στη δική μας επιτροπή να ξεκαθαρίσει ποια είναι η σωστή άποψη, ποια είναι η σωστή ανάλυση των στοιχείων. Το θέμα του καδμίου ήταν κάτι πολύ σοβαρό, το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Οι εμπειρογνώμονες είπαν ότι μία φορά συνέβη. Ήταν μία ακμή, αν θέλετε, στη γραφική παράσταση της μόλυνσης. Θέλω η γραμματεία να μας δώσει κάποιο προσανατολισμό. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να μην κοχλάζει το θέμα συνεχώς, δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει καλό ούτε στον αναφέροντα που σύρθηκε μέχρι εδώ να δώσει στοιχεία και θα φύγει χωρίς να βλέπει κάποιο τέρμα φως στην άκρη του τούνελ. Πρέπει να το λύσουμε το θέμα για την οικογένεια Μπρέναν, διότι αυτοί υπέφεραν επί μακρόν. Λοιπόν, είναι ανοιχτό θέμα. Εμείς, η Επιτροπή Αναφορών, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να μην σιγοβράζει το θέμα χωρίς ε, καμία λύση, να μην κοχλάζει. First, there is a basic principle. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Μπουστινάρου, έχουμε μια βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο ρηπαίνων πληρώνει. Mm. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει ο ρηπαίνων να πληρώσει. Και αυτό που έχουμε εδώ, έχουμε μια σαφή υπόθεση ρήπανσης θεωρητικός δεν έχουμε ρηπαίνοντα. δοθισόν των αξιολογήσεων των πολύ αορίστων μας οδηγούν σε κάποια βάσιμα... Δεν έχουμε συγκεκριμένο ε, πόρισμα που μπορούμε να βγάλουμε. Στη σελίδα... Α, το σημείο 4. Στο έγγραφο που έχουμε παραλάβει. Στο φάκελό μας. Σε επιτροπή αναφορών. Τι λέει εκεί. Λέει ότι η EPA καταχώρησε αρμόδια αρχή βρήκε τρει παραβιάσει από τι πέντε. Διαπίστωσε πράγματι συνέβησαν τρει παραβιάσει από τι πέντε. Και τέσσερι, δύο περιπτώσει μη συμμόρφωση από τι τέσσερι που εικάζονται. Άρα το μισό. Άρα πώς να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει ρηπαντής όταν τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις έχουν ξεπεραστεί τα όρια από κάποιον που ρήπανε. Τελευταίο ερώτημα. Σταμάτησε η επιχείρηση δραστηριότητε. Αφού σταμάτησε τι δραστηριότητε, κατά θαυμαστό τρόπο ανέκαμψε το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει σε θαύματα ή χρειαζόμαστε κάποια επιστημονικά στοιχεία. Διότι αν δεν υπάρχει κάποιος που ρήπαινε, και έφνη στο περιβάλλον ανακάμπτει, ιδού το θαύμα. Άρα πρέπει να ζητήσουμε τον Άγιο Πατέρα να επισκεφθεί το μέρος και να το κηρύξει Άγιο Τόπο. Αστιάκι βέβαια, αλλά δεν είναι και ξεκάθαρα αστείο, 100% αστείο, διότι παίζουμε με αοριστολογίες και τύπους που καμιά φορά καλύπτουν δραματικές πτυχές και αυτό είναι απαράδεκτο. Αν υπήρξε ρήπανση. Οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας πρέπει να κατονομάσουν και να καταδικάσουν το ρήπαντι. Αν δεν υπάρχει ρήπανση. Τότε γιατί έχουμε ένα θαύμα μπροστά μας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, δεν κατονομάζεται κανέναν, δεν λέτε ε, υπήρξε παράβαση, ξέρουμε ποιος παραβίασε. Πληρώνει ο Ριπένον. Ναι, ιού. Αυτά που μας λέτε εδώ πέρα είναι θεωρούμε ίσως ενδεχομένως ασάφιες. Ας συζητήσουμε την τραγωδία που αντιμετωπίζει ο Γιωργός. Ποιος του πληρώνει αυτού νου. Τις παράπλευρες απώλειες, έτσι να το αποκαλέσουμε. Δεν μιλάμε για επιχείρηση του ΝΑΤΟ βέβαια, αλλά λόγω της κακής εφαρμογής των περιβαλλοντικών προδιαγραφών κάποιος την πλήρωσε. Και πλήρωσε πολύ ακριβά. Και εδώ εμείς δεχόμαστε αόριστα σε διατυπώσεις, άσχετες διατυπώσεις και από την Ιρλανδική Αρμόδια Αρχή, ούτως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να κατονομάσετε, να πείτε αυτό στέει, αυτό το έκανε. Και να πληρώσει. Και πότε θα πληρώσει άμα να πληρώσει. Έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται. Η αρμόδια Ιρλανδική αρχή εφάρμοσε σωστά τους κανόνες, προς, προσμέτρησε επακριβώς πόσο, τι ποσά έφτασε η ρήπανση, τι ποσοστά. Εγώ θα έλεγα, υποστηρίζω θερμά να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και είναι θεμελιώδες να πληρώσει εκείνος που ρήπανε. Ανεξάρτητα από το όνομα εκείνο που μόλυνε. Πρέπει να πληρώσει τελεία και παύλα. Ε, ευχαριστώ. Ορίστε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Κέλλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα ε, τα έγγραφα. Τα βρίσκω ενδιαφέροντα